Dear colleagues, best colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια που είμαι η συνάδελφος με την μεγαλύτερη θητεία στην Επιτροπή, έχω την τιμή να προεδρεύσω στην ε, συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα και, όπως μου είπε η γραμματεία, έχουμε απαρτία δηλαδή τουλάχιστον το 1 τέταρτο των μελών, 19 δηλαδή μέσα στην αίθουσα. Οπότε θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ε, εκλογή Προέδρου της Επιτροπής και θα ήθελα να ε, προσκαλέσω τους συναδέλφους να παρουσιάσουν υποψηφιότητες είτε εκ μέρους των πολιτικών ομάδων είτε με τη στήριξη τουλάχιστον τεσσάρων βουλευτών. Ποιος θέλει τον λόγο. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ τη ομάδας ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, θα ήθελα να παρουσιάσω την υποψηφιότητα για την Προεδρία αυτής της Επιτροπής ε, ενός προσώπου το οποίο γνωρίζουμε όλο παλιά. Πρόκειται για τον συνάδελφο Έλμαρ Μπρόκ. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Πρόεδρε επίσης να αναφερθεί στα πρακτικά και οι ευχαριστίες που θα ήθελα να απευθύνω προς τον μέχρι τούδε Πρόεδρο της Επιτροπής μας, κύριο Αλμπερτίνη. Θα ήθελα επίσης, Πρόεδρε, να προσθέσω και ένα στοιχείο το οποίο υποβάλλω στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Μπρόκ δεν μπορεί σήμερα το απόγευμα να βρεθεί ανάμεσά μας, διότι έχει υποχρεώσει υποχρεώσεις προς του Κοινοβουλίου στην ομάδα που ασχολείται με την σύνταξη της νέας διακυβερνητικής συνθήκης. Σας ε, μας έχει αποστείλει μια επιστολή λέγοντας ότι δεν ε, θα μπορέσει να παραστεί σήμερα μεταξύ μας και ότι δέχεται φυσικά υποψηφιότητα. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Να αναγνώσω λοιπόν ε, το μήνυμα επιστολή του κ. Μπρόκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ενημέρωσαν πως η πολιτική μου ομάδα σκοπεύει να με προτείνει ως πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή με τιμά. Και με ευχαρίστηση αποδέχομαι την ε, πρόταση αυτή. Όπως ξέρετε είμαι αυτή τη στιγμή ένας από τους τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την ε, διεθνή για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οπότε δεν είμαι σε θέση να παραστώ συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και στην διαδικασία εκλογής Προέδρου. Λυπούμε ιδιαίτερα, αλλά νομίζω πως ε, έχω ηθική υποχρέωση εναντί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστώ ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή. Ζητώ λοιπόν την κατανόηση της Επιτροπής και την στήριξή σας. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω πως ε, έχω εκπληρώσει όλες τις ε, υποχρεώσεις ε, του αξιώματος αυτού. Έλμαρ Μπρόκ. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μια ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Ίσως μπορείτε να μας απαντήσετε. Παραδοσιακά, όταν κάποιο αναλαμβάνει ερετό αξίωμα σε επιτροπή, ε, τον ρωτάμε αν έχει συμπληρώσει τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων. Δεν το αναφέρει αυτό ο ρητός και υπάρχουν νέοι κανόνες από την ε, πρώτη πρώτου. Εσείς θεωρείτε πως με την διατύπωση αυτή θεωρεί πως, ε, δηλώνει πως έχει εκπληρώσει υποχρέωση του. Κύριε Τάνοκ, σας ξαναδιαβάζω έχω ηθική υποχρέωση έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το εκπροσωπήσω κτλ. Και μετά έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα αυτό. Νομίζω είναι σαφές. Ναι. Οπότε, αφού δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, προτείνω να εκλέξουμε τον κύριο Μπρόκ διαβοής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω πως ως ε, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών θα θέλαμε να πούμε στον κύριο Μπρόκ πως ε, ελπίζουμε πως η εκλογή του πλέον θα προσδώσει μια ακόμη καλύτερη εικόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα έξω και πώς θα ενισχυθεί υπό την Προεδρία του η Επιτροπή. Και νομίζω πως όταν έρθει ο κύριος Μπρόκ αύριο θα ευχαριστήσει φαντάζομαι τον κύριο Αλμπερτίνη. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει πρόεδρος, θα εξακολουθήσω να προεδρεύω εγώ στην ε, εκλογή των τεσσάρων αντιπρόεδρων. Σας ενημερώνω λοιπόν πώς ε, μας ενημέρωσαν οι ομάδες πως οι υποψηφιότητες είναι ως εξής. Για την, ε, τον πρώτο αντιπρόεδρο Προβέρα, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Πάσκου, τρίτος ο κύριος Κόβατσε και τέταρτος ο κύριος Μάιερ. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Όχι. Κύριε Προβέρα, δέχεστε την υποψηφιότητά σας. Μάλιστα. Κύριε Πάσκου. Ναι, ευχαριστούμε. Κύριε Κόβατσεφ. και ο κύριος Μάιερ. Ο κύριος Μάιερ έχει γράψει το εξής. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραστώ σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών. Με συγχωρείτε, είχα προβλήματα στην πτήση μου. Μόλις με ενημέρωσαν πως θα πρέπει να είμαι παρόν είτε αυτοπροσώπος είτε μέσω γραπτής διαδικασίας. Με το email αυτό λοιπόν σας ενημερώνω πως είμαι υποψήφιος. Θα αποστείλω κατά τη διάρκεια του απογεύματος και επιστολή μέσω fax. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς. Κύριε Βόητας. Ε, ε, ε, κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους της GUE NGL θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που έστειλε με το γραπτό μήνυμα ο συνάδελφος ο κύριος Μέγερ λόγω της ευνηδιαστικής του αυτής δυσκολίας στο να είναι παρόν εδώ και εκ μέρους προσωπικά του συναδέλφου και της ομάδας αποδεχόμαστε, αποδέχεται την υποψηφιότητα και στηρίζουμε την πρόταση που διατυπώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Διαβοής. So that means that I can Άρα, καλή τύχη σε όλους στις νέες τους θέσεις. Τώρα θέλω ο κύριος Προβέρα να προεδρεύσει. So, thanks to everybody. Thank you. Everybody's invited to come here. Όλοι να έρθετε, όλοι. Κύριε Κόβατσεφ και εσείς. Mr. Tanok, I did. I did fill my declaration, Mr. Tanok. Εγώ έχω συμπληρώσει δήλωση οικονομικών συμφερόντων, κύριε Τάνοκ. That's perfect. Yes, dear colleague. I think that... Αγαπητέ συνάδελφε, πρέπει νομίζω πρώτα να καλωσορίσουμε ένα νέο μέλος. Τον πρώην πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον συνάδελφο Μπούζικ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Τώρα λέω να αρχίσουμε. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν προτείνονται αλλαγές. Άρα εγκρίνεται το σχέδιο. Καμία αντίρρηση. Όχι. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις του Προέδρου. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κώσιφο Παιδίου. Η συγγήτρια η κυρία Ουλρίκε Λούνατσεκ. Είναι δεύτερη εξέταση του σχεδίου και των τροπολογιών. Ναι, νέα τροπολογίες έχουν κατατεθεί και η συγγήτρια διαπραγματεύτηκε 18 συμβιβασμούς. Το λόγο έχει η συγγήτρια Ουλρίκε Λούνατσεκ για να παρουσιάσει τα θέματα που θέτουν οι τροπολογίες και οι συμβιβασμοί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Καλωσορίζω και το νέο Προεδρείο της Επιτροπής με τους νέους Πρόεδρους και Αντιπροέδρους. Τώρα, όσον αφορά την έκθεσή μου, είχα μια συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές την προηγούμενη εβδομάδα και συμφωνήσαμε σε αρκετά σημεία. Πριν ξεκινήσω και πριν μπω στην ουσία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες και ειδικά όσον αφορά το κοσφοπέδιο, ξέρετε, η κατάσταση και η στάση στο κοσφοπέδιο ε, εξακολουθεί να διαφέρει και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες ε, για να δούμε βεβαίω μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σε κάποια δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Σε σχέση με την ε, τελευταία έκθεση τώρα πριν από 1,5 έτος έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Κάποια άλλα όχι. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει και το λέμε αυτό στο ψήφισμα στην ε, Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου του 2010, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχαμε ένα ψήφισμα το οποίο αποτέλεσε την αρχή διαλόγου μεταξύ ε, Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Μέχρι στιγμής είχαμε νέα συνεδριάσεις, ε, συναντήσεις τέτοιες, χωρίς βεβαίως να έχουμε όλα τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θα αναμέναμε, αλλά τουλάχιστον ο διάλογος αυτός ξεκίνησε και για πρώτη φορά εκπρόσωποι των δύο κρατών, των δύο κυβερνήσεων ε, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, κάτι το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος στις σχέσεις ε, των δύο κρατών. Αλλά γεγονότα. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα η Επίτροπος Μάλμστρομ πήγε στην Πριστίνα και ξεκίνησε τον διάλογο για τη Βίζα, κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει πριν από 1,5 έτος ως κοινοβούλιο. Πέρασε πολύ καιρός, αλλά επιτέλους ξεκίνησε και βεβαίως ε, και αυτό το σχολιάζουμε θετικά στην έκθεση. Επίσης, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2010, όταν 69 μέλη του ΟΗΕ είχαν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο, έχουμε φτάσει τώρα στα 85. Εξακολουθούν να μην είναι τα μισά μέλη του ΟΗΕ, αλλά είναι μια σημαντική αύξηση. Και αυτό άρα με οδηγεί στο επίμαχο σημείο μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας εδώ μέσα και στην έκθεση αυτή όπως και στην προηγούμενη έκθεση επαναλαμβάνω και ελπίζω να το πει η πλειοψηφία πως καλωσορίζουμε, εγώ καλωσορίζω, θα θέλαμε τα πέντε μέλη, κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο να το κάνουν. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουμε την μεγαλύτερη πολιτική μη στρατιωτική αποστολή της Ένωσης ε, στο Κοσμοπέδιο. Έχουμε πολύ προσωπικό ε, από διεθνείς οργανισμούς, ε, πολλά έργα της Κομισιόν και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στάση ενωμένη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αντιπροσωπείες εκείνες των κρατών μελών που δεν έχουν αναγνωρίσει αλλά έχουν γραφεία συνδέσμου στην Πριστίνα Κάτι το οποίο νομίζω δίνει μια ένδειξη πρόοδου, πιθανής πρόοδου. Κάποια άλλα γεγονότα που αναφέρω στην έκθεσή μου είναι πως είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένου και του χθεσινού ε, δημοψηφίσματος στην ε, Κροατία το οποίο είχε ένα αποτέλεσμα θετικό με βρισφία δύο τρίτων ε, είναι πως η προοπτική που υποσχεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη το 2003 εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτό ισχύει και για το κοσμοπέδιο και το τονίζω στην έκθεσή μου. Ανέφερα ήδη τη σημασία του διαλόγου με το Βελιγράδι, ανέφερα τη σημασία του να ξεκινήσει ο διάλογος της Βίζας για να καταργηθεί η αίσθηση της απομόνωσης που έχουν οι νέοι του κοσφοπεδίου σε σύγκριση με τους πολίτες όλων των γειτονικών χωρών που μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ενώ αυτοί δεν μπορούν. Και ε, τους δημιουργείται η αίσθηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει στα σοβαρά αυτή την προοπτική. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκίνησε ο διάλογος για την Βίζα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε έναν οδικό χάρτη και μετά βεβαίως επαφείται στην ε, κυβέρνηση Κοσφοπεδίου να εφαρμόσει τα σχετικά βήματα. Κατόπιν στην έκθεση αναφέρομαι και στους προβληματικούς τομείς στο ίδιο το κοσφοπέδιο. Είχαμε σοβαρές παρατυπίες στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Αρκετοί συνάδελφοι είχαν πάει εκεί ως παρατηρητές των εκλογών και ζητώ στην έκθεση εγώ να τιμωρηθούν γρήγορα και επαρκώς όσοι διέπραξαν απάτη ειδικά στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα. Γιατί πρέπει να δείξουμε στους πολίτες κοσφοπεδίου πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά σε εκλογές. Επίσης ε, ζητώ και από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν γρήγορα στις αλλαγές του συντάγματο και του εκλογικού νόμου οι οποίες είναι απαραίτητε για ε, να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές και να μην υπάρχουν προβλήματα με τα ψηφοδέλτια και τη διεξαγωγή της ψηφοφορία για να έχουμε σωστές εκλογές την επόμενη φορά. Το ζήτημα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος είναι κάτι το οποίο απασχολεί την EULEX και την έκθεσή μου, το κράτος, η αποστολή αυτή που αφορά το κράτος δικαίου, η EULEX έχει ειδικού τομεί, ασχολείται με τα τελωνία, την αστυνομία και θεωρούν ήδη πως μπορούν να μειώσουν το προσωπικό γιατί έχει υπάρξει πρόοδος τόπου. Εκεί όπου πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα είναι στη διαφορά υψηλού επίπεδου και στο οργανωμένο έγκλημα, στην προστασία των μαρτύρων και στις δύο πλευρές και στο κοσφοπέδιο που πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για την προστασία των μαρτύρων αλλά και ε, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην EULEX θα πρέπει να είναι διαθέσιμα να δεχτούν στις χώρες, ε, στις χώρες τους ε, μάρτυρες. Επίσης ε, υπάρχει το ζήτημα το οποίο φαίνεται πάρα πολύ βέβαια στα μέσα μαζικής είτε η τεταμένη κατάσταση στο βορρά. Εκεί πέρα ζητάω να φύγουν τα οδοφράγματα, και ζητάω από τη σερβική κυβέρνηση να διαλύσει τις παράλληλες δομές ε, που είναι η βάση των διαμαρτυριών. Επίσης ξεκαθαρίζω πως ε, η απόσχηση δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. I think uh, Και είναι απαραίτητο, νομίζω, και η κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου θα πρέπει να πείσει τον σερβικό πληθυσμό όπως είναι και δική τους η χώρα και να κάνει ένα πρόγραμμα σχετικά και βεβαίως να φύγουν τα οδοφράγματα και να διαλυθούν οι παράλληλες δομές των Σέρβων. Αυτό το οποίο καλωσορίζω είναι η αυξημένη εμπλοκή της ε, σερβικής κοινότητας, ειδικά νοτίως του Ήμπαρ ε, και όσον αφορά την προστασία της ε, πολιτικής κληρονομιάς. Υπάρχουν και κάποιες θετικές πτυχές λοιπόν, τις οποίες θα ήθελα να τονίσω. Ε, όσον αφορά τη χώρα αυτή των Δυτικών Βαλκανίων. Καλωσορίζω επίσης ε, την σύσταση της ειδική ερευνητική ομάδας ε, της EULEX που ενδιαφέρει πολλούς βουλευτές και αφορά την διερεύνηση της έκθεσης Μάρτη που μιλούσε για εμπόριο οργάνων ήδη στον καιρό του πολέμου και μετά αλλά και πιο πρόσφατα έχει συσταθεί αυτή η ομάδα, βασίζεται εδώ στις Βρυξέλλες, ε, εδώ έχει την έδρα της και ελπίζω σύντομα να έχει αποτελέσματα. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την ελευθερία των ΜΜΕ, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις ε, στο κοσφοπέδιο που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις αναφέρω στην έκθεσή μου, ειδικά όσον αφορά τα ανεξάρτητα ΜΜΕ που αποτελούν βεβαίω θεμέλιο λίθου τη δημοκρατία. Όχι μόνο στο κοσφοπέδιο και αλλού στα Δυτικά Βαλκάνια και στι χώρε μα, όπω ξέρουμε και συζητάμε συχνά. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε επίσης είναι να εστιάσει περισσότερο η κυβέρνηση στην κατάργηση των διακρίσεων, είτε μιλάμε για τι γυναίκε είτε μιλάμε για διάκριση με βάση την θρησκεία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά κυρίως για διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Μίλησα ήδη για τους Σέρβους, αλλά και Ρώμα κλπ. Αυτό το οποίο βρήκα λοιπόν θετικό ήταν πως ε, έχει υπάρξει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν. Υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα παρόλα αυτά. Έχουμε, είχαμε προβλήματα γενικώ με την οικονομία γιατί ε, υπάρχουν ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, μια πολιτική βιώσιμη δημοσιονομική η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι το πολύ σημαντικό και έχει ελλείψεις. Some, there uh, Υπάρχουν κάποιες ε, θετικές εξελίξεις, αλλά το βασικό πρόβλημα υπάρχει είναι η παραγωγή ενέργειας. Υπάρχει το πρόβλημα δύο ε, εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, το Κόσοβο Α και το κόσμο Β που ρηπαίνουν. Το Κόσοβο Α θα πρέπει να κλείσει το μότρο δυνατόν και το Κόσοβο Β και αυτό επίσης. Αυτό για το οποίο λυπάμαι είναι πως δεν έχουν γίνει, γίνει έρευνες για να δούμε το τι μπορεί να γίνει αντί για αντί για αυτούς τους ε, σταθμούς. Ε, Γενικώ λοιπόν να πω πως γνωρίζω πως ε, στο Κοινοβούλιο έχουμε και βουλευτές που ακόμα δεν συμφωνούν με την ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου αλλά σας ζητώ να σκεφτείτε πως η χώρα αυτή είναι μέρος της πολιτικής διεύρυνσης, μέλος της διαδικασίας της Θεσσαλονίκης και πρέπει να προωθήσουμε την ευημερία των κατοίκων αυτής της χώρας και ελπίζω να στηρίξετε και τις συμβαστικές προτάσεις που έχουμε εδώ πέρα γιατί όπως είπα είχαμε πολύ καλή συνεργασία με όλες τις ομάδες του Κοινοβούλου. Ευχαριστώ. Thank you. And... Ευχαριστώ. Τέσσερις συναδελφοί έχουν ζητήσει το λόγο. Προηγουμένως όμως να καλωσορίσω τον Υπουργό Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος ε, του Κοσυποπεδίου. Ο σκιώδης ηγητής κύριος Πόσελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ για την ισορροπημένη αυτή έκθεση και είπα πως η έκθεση αυτή δεν θα έπρεπε καν να αλλάξει σε τίποτα. Και το ότι υπάρχουν 209 τροπολογίες και δικές μου και της κυρίας Λούνατσεκ οφείλεται στα πάρα πολλά μυστικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θα μπορούσαμε να την ψηφίσουμε στην αρχική της μορφή. Τώρα τέλος πάντων έχουμε 209 τροπολογίες. Χαίρομαι για την καλή συνεργασία που είχαμε με όλους τους κοιόδης για να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες που καθιστούν τις περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές περιτές. Εάν μου επιτρέπετε τώρα να αναφέρω κάποια πράγματα, να προσπαθήσω να αξιολογήσω κάπως πολιτικά τις τροπολογίες. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που προσπαθούν ξανά να θίξουν το ζήτημα του καθεστώτος. Και πρέπει να πω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με πλειοψηφία τριών τετάρτων ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας του κοσφοπεδίου είπε με πλειοψηφία τριών τετάρτων πως δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε το ζήτημα του καθεστώτος και θέλω να πω πως κάθε φορά που θα συζητάμε το κοσφοπέδιο έχουμε ξανά τις ίδιες τροπολογίες για το καθεστώς, για τη διατύπωση, το εάν είναι δημοκρατία, το εάν έχει πολίτες και να ψηφίζουμε ξανά τα ίδια πράγματα είναι ε, και ενοχλητικό. Σέβομαι το οτι 5 πέντε κράτη-μέλη από τα 27 έχουν μια διαφορετική θέση. Αλλά 22 κράτη-μέλη έχουν λύσει οριστικά μέσω της αναγνώρισης το ζήτημα του καθιστότος. Το ίδιο ισχύει για 85 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Όλες οι χώρες των G7 όλες οι γειτονικέ χώρες του Κοσφοπεδίου, οπότε δεν έχει νόημα, θεωρώ, να συζητάμε ξανά και ξανά το ζήτημα του καθιστώτος. Και το λέω ξεκάθαρα, το σέβομαι να έχει μειοψηφία άλλη γνώμη, αλλά δεν μπορεί η πλειοψηφία να απαιτεί η μειοψηφία να την ακολουθήσει. Γι' αυτό δεν λέμε στο κείμενο αυτό, ε, δεν λέμε κι εμείς πως απαιτούμε από τα πέντε κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν, όχι ζητάμε γενικά για να υπάρχει μια ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό θα διευκολύνει και τη δουλειά της EULEX. Είναι ήδη προβληματικό το ότι για ένα τόσο θεμελιώδες συζήτημα δεν έχουμε συμφωνήσει μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια δυναμία της εξωτερικής πολιτικής την οποία πρέπει να αποδεχτούμε γιατί βεβαίως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αλλά μετά αποδεχτείτε σας παρακαλώ και αυτά τα οποία λέει η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Ε, είναι επικίνδυνο να ανοίγουμε κάθε φορά το θέμα του καθεστώτος. Το ίδιο και για τον διχασμό του κοσφοπεδίου. Εμφανίζεται ξανά και ξανά αγαπητοί φίλοι, ως κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλά νομίζω την περιοχή, θα ήθελα να σας αποτρέψω να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τι συνέπειες θα έχει αυτό μετά. Γιατί τότε θα έχουμε φύγει για πρώτη φορά από την αρχή ότι έχουμε ως βάση τα σύνορα της παλαιάς Ιουγκοσλαβίας. Και μετά τι θα γίνει με τους Αλβανούς Σερβίας, το Πρέσεβο, τι θα γίνει στην ε, Πουγουδουμού και εκεί πέρα πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα, στο Σαντζάκι του Νοβι, Νόβι Παζάρ, οπότε σας παρακαλώ μην ανοίγεται αυτό το θέμα. Οπότε, το βασικό ζήτημα είναι η EULEX. Η μεγαλύτερη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλές απαιτήσει. Έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά έχει και πολλές προσδοκίες τις οποίες απογοήτευσε και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να σταθούμε επικριτικά η EULEX θα πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική σε ολόκληρη την επικράτεια του πεδίου και το να την στηρίξουμε είναι αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, μέρος αποστολής του ως Δημοσιονομική Αρχή δύο ακόμα σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι ο διάλογος για τη βίζα. Δεν είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να κάνει απελευθερωτικό πόλεμο και μετά οι άνθρωποι τους οποίους απελευθέρωσε να μένουν περίκλειστοι στη χώρα τους και όλες οι γειτονικέ χώρες να έχουν ε, ε απαλλαγή από τη βίζα. Πώς να νιώθουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία ο διάλογος για τη βίζα και κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε, η εμπορική συμφωνία, η χώρα αυτή έχει πολύ νεανικό πληθυσμό, ο οποίος χρειάζεται θέσεις εργασίας, αλλιώς δεν θα έχουμε σταθερότητα. Γι' αυτό χρειάζεται εμπορική συμφωνία με την Ένωση, γι' αυτό χρειάζεται ασφάλεια δικαίου, προώθηση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη εναλλακτική ενέργεια Εκεί πέρα συμφωνώ με την κυρία Λούνατσεκ. Είναι κάτι το οποίο έχει νομίζω πολλές ικανότητες σε αυτή τη χώρα. Τέλος θα ήθελα να πω, τα ζητήματα των μειονοτήτων στη χώρα έχουν ρυθμιστεί θαυμάσια με βάση το σχέδιο Αχτισάρη και θα πρέπει επιτέλους να δεχτούμε πως το 6% των Σέρβων που ζουν στο κοσμοπέδιο, από αυτό το 6%, 4% έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε αυτό το νέο κράτος, αυτοί που ζουν στο Νότο και είναι το 1 τρίτο, δηλαδή μια πολύ μικρή πλειοψηφία των Σέρβων, στο Βορρά που δημιουργούν δυσκολίες και μέσω των παράλληλων αυτών δομών. Γι' αυτό και η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών είπαν ξεκάθαρα πως οι παράλληλες αυτές δομές πρέπει να εξαφανιστούν και εάν δεν διαλυθούν, το λέω αυτό ξεκάθαρο, δεν θα υπάρξει και καθιστός υποψηφιότητα για την Σερβία, το οποίο επί της αρχής εγώ ε, θα ήθελα βεβαίω να υποστηρίξω, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να διαλυθούν αυτέ οι παράλληλε δομέ του κοσφοπεδίου. Ευχαριστούμε. Δεύτερο σκιώδη, ο κύριο Παντζέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι κατά τη συντομότερο. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Λούνατσεκ, αλλά και φυσικά όλου του σκιώδη ηγητέ με τους οποίους είχαμε επικοδομητική συνεργασία και που κατέληξε στους πολλούς συμβασμούς που έχετε αναχείρας ε, συμβασμούς, ο οποίους ε, υποστηρίζω και θεωρώ ότι είναι απόλυτα ισορροπημένοι. Πέραν αυτών των ε, συμβαστικών προτάσεων έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες που φροντίζουν να αντιμετωπίσουν διάφορες προβληματικές που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες π.χ η ανάγκη ενίσχυσης περαιτέρω του κράτους δικαίου και το δικαστικό σύστημα και να καταστήσουμε το εκλογικό σύστημα πιο διαφανές ε, να διασφαλίσουμε τον απαραίτητο συντονισμό και την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των ε, Υπουργείων και μια μεγαλύτερη τεχνική στήριξη στις ε, δομές συντονισμού. Τέλος, σε σχέση με το EULEX, να πω ότι αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε διάφορες διαφορετικές ελλείψεις όπως η έλλειψη <clears throat> ε, ελέγχου και να εξετάσουμε διάφορες πτυχές διαχείρισης και προγραμματισμού προκειμένου να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές που τουλάχιστον εγώ κρίνω απαραίτητες. Πάντως να ευχαριστώ για μια ακόμα φορά την εισηγήτρια για την εργασία της. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν είναι διόλου απλό, αλλά είμαι πεπισμένος ότι δούλεψε αποτελεσματικά και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε ενωμένοι για την στήριξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής, ο κ. Κάτσιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ την κυρία εισηγήτρια, κυρία Λούνα Τσεκ, που δεν είναι μόνο ενθουσιώδης ε, για το θέμα αυτό, αλλά και πραγματικά ε, μας ε, προχωρεί το ζήτημα του Κοσμοποδίου με τον κατάλληλο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω, θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο διάλογος να ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ζήτημα πάρα πολύ συγκινησιακό και φορτισμένο συγκινησιακά θέμα, όπως αυτό της ε, ε, δικαστικής συνεργασίας και θα υπάρξουν μέσω αυτού του διαλόγου η εξίσωση των, του πληθυσμού του Κωσυφοπαιδίου με τους υπόλοιπους ε, της περιοχής. Θα ευχαριστήσω λοιπόν την Κομισιόν που ξεκίνησε αυτό το διάλογο. Από την άλλη πλευρά όμως Χρειάζεται να αναφέρω πως οι πρόσφατη εξελίξεις στο Κοσμοπέδιο και ιδιαίτερα οι διάφορες διαδηλώσεις που οργάνωσε ο Άρντεχουρτ και το κόμμα του είναι μια, ε, κάτι το αρνητικό, ένα αρνητικό μήνυμα για μας. Είναι λυπερό που το, ε, ε, το Βελιγράδι δέχθηκε να αφήσει την ελευθερή κυκλοφορία των προσώπων και ξαφνικά συνέβη κάτι το αρνητικό από πλευρά ε, κοσμοπεδίου. Η λαϊκιστική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και πιστεύω ότι το κοινό στο κοσμοπέδιο θα πρέπει να ε, ε, ασχοληθεί με τις προκλήσεις αυτές του Κούρτη στα σοβαρά πραγματικά θα οδηγήσει το κοσμοπέδιο σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και Επίσης ε, να αναφέρω πως ε, θα πρέπει να συγχαρούμε για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις και την σημερινή αγγελία της κυρίας Ταχύρη η οποία δήλωσε πως ε, υπάρχει πρόοδος στο ζήτημα της ονομασίας το όνομα με το οποίο θα συμμετέχει το κοσμοπέδιο στα διάφορα διεθνή φόρα το κοσμοπέδιο στην... χωρίς υποσημειώσεις είναι μια πολύ καλή πρόταση. Την υποστηρίζει το κοσμοπέδιο και θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Βελιγράδι. Αυτό θα δημιουργήσει λοιπόν μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλύτερο κλίμα και δυνατότητες για αμοιβαίο συντονισμό και αμοιβαία συνεργασία και θα προσεγγίσει όχι μόνο τις δύο τις πλευράς αλλά όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και δει ε, όσες δεν έχουν ε, αναγνωρίσει ακόμα το κοσμοπέδιο. Και μια τελευταία ερώτηση. Ελπίζω πως σύντομα θα είμαστε σε θέση να οργανώσουμε ένα hearing για με ακρόαση με τον νέο επικεφαλής της Επισοφίας του Κοσμοπεδίου. Θα είναι εξαιρετική ευκαιρία για να συνεχίσουμε την συζητήση μας επί του Κοσμοπεδίου ναι, άκουσα, άκουσα τι είπατε, οι διερμηνείς όμως δεν άκουσαν. Ναι, ξέρουμε ότι καθυστέρησε λίγο. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε έναν νέο επικεφαλής της Ευσοπίας, ο οποίος ε, δεν θα χρειαστεί να μετακινηθεί και να λάβει υπουργική θέση. Αυτό νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικό για το για την σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Η ομάδα μου υποστηρίζει την έκθεση Λούνατζερ και φυσικά εύχεται για την ειρήνευση του Κωσυφοπεδίου αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία είναι η συγκολητική ουσία που συνδέει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και διασφαλίζει την ένωμη τάξη, την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, την ελευθεροτυπία κλπ. Αν αυτή η συγκολητική ουσία πάψει να υπάρχει, τότε θα υπάρξει πραγματικός κίνδυνος αποσταθεροποίησης και από τις δύο πλευρές της διαμάχης του Κωσυφοπεδίου. Φυσικά προτεραιότητα πρέπει να είναι η στήριξη της Γιούλεξ από την Ένωση και στην καταπολέμησή της της διαφθοράς και δωροδοκίας και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της εξάρτησης του Κωσυφοπεδίου από τη Δυτική Ευρωπαϊκή Ιδίως Βοήθεια. Η Λέβη Άστον ανέλαβε διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνης και ελπίζουμε τελικά να επιτευχθεί ευημερία και για τις δύο πλευρές αν και η μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να συζητηθεί κάποτε διεθνώς. Η δήλωση του κυρίου Πόσελτ ότι μόνο μία μικρή μειονότητα Σέρβων ε, δημιουργεί τις ταραχές νομίζω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι μεγάλη πλειοψηφία των Σέρβων δεν δέχονται την κυριαρχία της Πριστίνης. Γι' αυτό φοβούμε ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της αποκοπής του κοσυφοπεδίου δεν θα του επιτρέψουν να μπει ούτε στην Ένωση ούτε πουθενάλλου. Η μη αναγνώριση από ορισμένε χώρες μέλη και χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπως η Κίνα και η Ρωσία δεν ξέρω αν θα αλλάξουν στάση. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Αλλιώς τα προβλήματα θα συνεχίσουν και το κόστος θα είναι τεράστιο για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και φορολογούμενες. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κούκεν, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω το ψήφισμα που θα δεχτούμε τελικά να είναι ισορροπημένο και να αναφέρεται στις τα πραγματικά προβλήματα του κοσυφοπεδίου. Το σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας είναι καλό και εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία της εισηγήτριας που επεξεργάστηκε τους συμβιβασμούς. Τέσσερις δηλώσεις έχω να κάνω σχόλια. Πρώτον, για το διάλογο για τις θεωρήσεις που ανέλαβε η Επίτροπος Βάλστρομ. Ο διάλογος αυτός θα είναι δοκιμή για το κοσυφοπαίδιο. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές όπως κάναμε προηγουμένως και με άλλες χώρες της περιοχής. Κατάλαβα ότι η έκθεση αυτή δεν αναφέρει το σχεδιασμό δημοψηφισμάτων στη Σερβία για το Κωσυφοπαίδιο γιατί αυτό θα δυσκόλευε τα πράγματα. Με χαρά σημειώνω ότι η Σέρβη πολιτική δεν είναι υπέρ των δημοψηφισμάτων και ελπίζω τελικά να αποσύρουν την ε, υποστήριξή τους παραλλήλων πολιτικών δομών στο βορρά του Κωσυφοπεδίου. Η Γιούλεξ και η δουλειά της στο Κωσυφοπαίδιο πρέπει να επανεκτιμηθεί με βάση των αποτελεσμάτων που έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πρέπει βέβαια να έχουμε πληροφόρηση για τα σχέδια αναδόμησης της αποστολής αυτής και να δοθεί ιδέουσα σημασία στο θέμα. Για την ενέργεια σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι θα αυξηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του κοσυφοπεδίου με τον χρόνο, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία από τους υπάρχοντες σταθμούς. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι οι νέες πηγές ενεργείας δεν έχουν προσεχθεί εκεί και τώρα μάθαμε ότι μπορεί να ξανανοίξει ο σταθμός Α2 που είναι απαρχαιωμένος και δεν έχει εξυγχρονιστεί τα τελευταία 11 χρόνια. Τέλος, οι διαδηλώσεις με σύνθημα για την αμοιβαιότητα των εμπορικών σχέσεων Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Δικαίωμά είναι μεν οργανώνουν διαδηλώσεις, αλλά πρέπει να σέβονται αυστηρά όλους τους κανόνες για να μην δυσκολεύουν την κατάσταση χωρίς να χρειάζεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα συνάδελφοι έχω πέντε ακόμη ομιλητές και σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Η κυρία Αμονήθη πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδης ηγητές. Θα ε, να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν θεωρώ ότι μια, ε, μια επικοδομητική στάση αλλά διαφοροποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει θετικότατα στην στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτή η προσέγγιση είναι ε, αυτό που επέτρεψε σε συνεδριάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ε, χώρες των Βαλκανίων, η πρώτη υπό Ισπανική Προεδρία 2010 και την ομόφωνη θέση που στηρίξαμε στον, ε, στηρίξαν στα Ηνωμένα Έθνη για τη Σερβία, τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τον διάλογο με την Πρίστινα. Πρέπει να αποφύγουμε να διχαστούμε και να χωριστούμε σε θέματα όπως αυτό. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην χώρα αυτή κλπ. Θέλω να κάνω όμω και κάποιε άλλε σκέψει. Καταρχήν η σημασία του να εγκριθεί η τροπολογία 2 προκειμένου να μην εμπλακούμε στο θέμα του ονόματο του Κοσμοπεδίου. Θα πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε στις 244 συγγνώμη, του απόφαση των ΗΠΑ και όλε οι αναφορέ που γίνονται στο Κοσμοπέδιο ε, υπό την Γίνονται χθε υπό την επιφύλαξη του καθεστώτος του 20 πεδίου. Δεύτερον, στην εμβαστική πρόταση 1 δεν μπορούμε να ζητήσουμε την υποχρεωτική ε, αποδοχή της έγκρισης ε, τη αναγνώριση του 20 Υπάρχει ένα συμβασμό στον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα μειονοτήτων ε, πλειοψηφιών, πρόκειται για ένα θέμα κυριαρχίας ενός κράτους να παρατηρήσω επίσης ε, πως θα πρέπει να γνωρίσουμε τις ε, προσπάθειες ε, που έχουν καταβληθεί από πλευράς Πρόεδρου Τάντιτς στις 29 Νοεμβρίου κάλεσε να αποσυρθούν τα οδοφράγματα και στις και τον Ιούλιο είχε ζητήσει να στους Σέρβους να κρατήσουν την ψυχραιμία του Στην παράγραφο 7 λοιπόν τη συμβαστική πρόταση 6 αναφέρονται statements στο πληθυντικό και όχι statement διότι ο πρόεδρο Τάτζιτ ε, έχει κάνει διάφορε δηλώσει, υπέρ τη ε, ηρεμία και τη ψυχραιμία που πρέπει να επιδείξουν οι πληθυσμοί. Ευχαριστώ όλου του εισηγητέ και σκιώδει εισηγητέ. Ευχαριστώ κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για τον επαγγελματισμό της ε, και τη συγχαίρω για την έκθεσή της. Συμφωνώ με όλους πως ε, πραγματι υπάρχει πρόοδος μετά το χθεσινό δημοψήφισμα στην Κροατία όπου δύο τρίτα των ψηφοφόρων αποφάσισαν να υπερψηφίσουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σωστό να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ευρωπαϊκή προοπτική και σε άλλες ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω πως πρέπει να στηρίξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες που προσθέτουν στην έκθεση, ειδικά όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, ε, καθώς αυτό αφορά πραγματικά τον ε, κόσμο, τους ανθρώπους. Δεν θα αναφέρω τώρα άλλα επιχειρήματα, απλά θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Η συγγήτρια ανέφερε νέα συναντήσεις που είχαν γίνει στο πλαίσιο του ε, διαλόγου. Άλλα έγγραφα νομίζω αναφέρουν 8 ή 5. Νομίζω πρέπει να καταλήξουμε σε έναν αριθμό. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και οι στην συνάδελφοι, να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές που δούλεψαν ε, προκειμένου να συντάξουν την έκθεση αυτή η οποία είναι πολύ καλή, πολύ απόλυτα κατανοητή, ε, επικοδομητική. Δεν ε, μιλάει μόνο για τα προβλήματα, αλλά προσπαθεί να εντοπίσει ποιοι είναι οι τομείς όπου έχει υπάρξει απαιτείται πρόοδος ε, στο πεδίο, ε, ε, Που κινούμε το ζήτημα της Σερβίας που προετοιμάζεται θα στείλουμε ένα ορθό μήνυμα προς την περιοχή. Θα ήθελα να τονίσω όμως πως και επιθυμώ να εργαστούμε λίγο παραπάνω στον οικονομικό κλάδο, να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, καταπολέμηση της ε, διαφθοράς ε, και της παράλληλης οικονομίας, της παραοικονομίας και όλα τα ζητήματα που αφορούν της τι τις μεταφορές, τα δίκτυα κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα προορατικό ρόλο για να βοηθήσουμε το οικοσοπαίδιο προκειμένου να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και σε θέματα γεωργίας, ζητήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ε, το Κοσμοπέδιο μπορεί να καταστεί μια χώρα η οποία θα παρέχει, θα εξάγει ε, ηλεκτρική ενέργεια. Ξέρετε ότι και υπό την προηγούμενη αποστολή της ΑΝΜΙΚ δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος για θέματα οικονομίας. Ε, καλωσορίζω τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Αντιπροσωπής του Κωσοπέδιου στις ε, Βρυξέλλες αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να δραματίσουμε έναν πιο ενεργό ρόλο στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιαννάκου, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ε, υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το Κόσοβο ε, και ότι οι πέντε χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει και δεν βρίσκουν λόγους ακόμη να αναγνωρίσουν ε, ε, αυτή την πραγματικότητα. Θέλω να σημειώσω όμως το θετικό στοιχείο που έγινε, η πρόοδος δηλαδή, ότι έχουν αρχίσει συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί χωρίς αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, δια της επιβολής εκ των έξω, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει οτιδήποτε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας φυσικά αυτά που έγιναν στις εκλογές, όχι μόνο ώστε να μην επαναληφθούν, αλλά ώστε και να κρατηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια και ανάμεσα στις διάφορες εκλογές. Ε, και εκεί εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιη ότι η κατάσταση είναι τόσο ευτυχής όσο περιγράφεται. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ χειρότερη ε, και ότι το εσωτερικό, η εσωτερική κατάσταση δεν ανταποκρίνεται ε, σε αυτά που ενδιαφέρουν εμάς και θέλουμε να εμφανίζουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο έντονο τρόπο να παρέμβει στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, last speaker. Ε, hvala lepa, ja, hvala lepa predsedujoči. Tudi jaz bi se najprej um, pridružila vsem zahvalam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία αλλά και για την προσπάθεια που έχει καταβάλει προκειμένου το Κοσμοπέδιο να ε, ενταχθεί στην, ε, κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εντάσεις ε, που προέκυψαν χθες μετά από τις εξελίξεις στην χώρα από το κόμμα Κούρπη δεν είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στο θετικό κλίμα στην περιοχή και ειδικά στις σχέσεις με την Σερβία. Ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι ξεκίνησε και ο διάλογος για το θέματα των προξενικών θεωρήσεων. Το, για το ζήτημα πάντα των θεωρήσεων χαίρομαι που υπάρχουν θερμικές εξέλιξεις για τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκονίων. Η διαδικασία αυτή είναι σίγουρα περίπλοκη, απαιτητική. Το κοσμοπέδιο θα πρέπει να πληρεί μια σειρά κριτηρίων, ειδικά σε θέματα κατά πολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και της διαφοράς. Πρέπει να οργανώσουν τα έλεγχο των συνόρων, το, να οργανώσουν την ασφάλειά της κλπ. Είναι κάτι το οποίο όμως το οποίο θα πρέπει να φέρει σε έζιο πέρας. πρέπει να φροντίσουμε η χώρα να μην απομονωθεί. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν ε, τον ε, Ιούλεξ. Χαίρομαι που πετύχαμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και καλωσορίζω επίσης ε, τον διορισμό του νέου επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοσμοπεδίου στις ε, Βρυξέλλες. Θα έχουμε αναφίβολα την ευκαιρία να τον συναντήσουμε πριν ξεκινήσει τις εργασίες του στο Κοσμοπέδιο. και κρίνουμε ότι θα μπορέσει να βρει τρόπους για να ξεπεράσει τις διαφορές που υπάρχουν αναφορικά με την αναγνώριση του κοσμοπεδίου. Παράλληλα θα ήθελα να σχολιάσω τα λεγόμενα της εισηγήτριας ε, σχετικά με την ε, κατάσταση στον ε, τομέα των μέσων ενημέρωσης και καλωσορίζω τις συμβαστικές τροπολογίες ε, που ζητούν την εφαρμογή των διεθνών στάνταρ για την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης διότι αυτό είναι και βάση για την δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με δέχεστε κιόλας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας. Ναι, νομίζω η πιο σημαντική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Επισκέφθηκα τα Δυτικά Βαλκάνια πριν από δύο μήνες. Συγχαίρω την κυρία Λούνατσεκ και όλους τους σκιώδες ηγητές για την πολύ καλή αυτή έκθεση και συμφωνούμε στο περισσότερο σημείο. Μία διαφωνία έχουμε που έχει σημασία βεβαίως, ε, την αναγνώριση του κοσφοπεδίου. Τα υπόλοιπα το ξέρουμε, όσο έχουμε την ίδια άποψη. Δημοκρατία, ελεύθερα μηνιαία, οικονομία της αγοράς κτλ. Αλλά να τονίσω ένα πράγμα. Τα σημαντικότερα προβλήματα, εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις για μια καλύτερη συμβατότητα του κοσφοπεδίου με την Ένωση βεβαίως ε, βρίσκονται στις διμερείς σχέσεις με τη Σερβία και από την άλλη όλα τα επιτεύγματα και η έγκριση, αν θέλετε, η δική μας για τη μελλοντική συμμετοχή της Σερβίας να εξαρτάται από τις σχέσεις της Σερβίας με το Κοσφοπέδιο. Οπότε νομίζω πως η δική μας υποχρέωση σήμερα είναι να βελτιώσουμε την συνεργασία των δύο αυτών χωρών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα μπρος στην περιοχή αυτή χωρίς συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Και μπορούμε να βοηθήσουμε και τις δύο χώρες. Και τα Δυτικά Βαλκάνια. Όσο νομίζω ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής ε, στα σημαντικότερα ζητήματα μεταξύ των ε, δύο χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής Σεφλίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Μπούζεκ. Πράγματι το θέμα της Σερβίας παίζει ε, σημαντικό ρόλο και πράγματι η σερβική μειονότητα ε, του παιδίου γιατί συμφωνώ πλήρως με τον στόχο της ε, ένταξης ε, που αναφέρεται και πρέπει να ενταχθεί η σερβική μειονότητα στο κοσμοπέδιο πλήρως στις πολιτικές και λοιπές δομές αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως πως δεν θα είναι απλή αυτή η διαδικασία. Μάλιστα να το δούμε σε ένα ιστορικό πλαίσιο η σερβική μειονότητα στο κοσμοπέδιο είχε ένα προνομιούχο καθεστώς από τη στιγμή ε, στην οποία ενσωματώθηκε πρώτα στη Σερβία και μετά στη Ιουγκοσλαβία το κοσφοπέδιο. Το ότι έχασαν τώρα αυτό το καθεστώς θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να το αντιληφθούν και χρειάζεται και κάποια γενεοδορία από πλευράς πλειοψηφία. Οπότε η ένταξη αυτή, αν θέλετε, είναι μία υπόθεση που αφορά και τις δύο πλευρές και πάρα πολύ θα έλεγα και την πλειοψηφία. Και η διαδηλώσεις βεβαίως που έχουν υπάρξει δεν προσφέρουν καθόλου ασφάλεια στην ε, σερβική μειονότητα. Κύριε Λούνατσεκ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια των αδέλφων. Αλλά καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους όσοι με συνεχάρισαν και να ρυθμίσω μερικά πράγματα. Κύριε Πέτερ, είπατε ότι δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το 5, 7, 9 συναντήσει για το διάλογο. Ελέγξαμε την περίοδο εβδομάδα, 9 ήταν οι διάλογοι. Αυτή είναι λοιπόν η τελική εκδοχή. 9. Ευχαριστώ που διαβάσατε προσεκτικά το κείμενο και παρακολουθήσατε τις εξελίξει. Κάτι ακόμα, κύριε Γκόμες, αναφερθήκατε στο ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το αξιοπαίδιο μετά τις της οικονομίας. Χαίρομαι που το δηλώνετε. και επιθυμώ να έχουμε μια στήριξη στο Κοινοβούλιο για την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοσμοπέδιο. γιατί αυτό θα σημαίνει ότι υπάρχουν επίσημες σχέσεις, τυπικές σχέσεις μεταξύ των 27 και του Κοσμοπέδιου. Αυτό θα μας βοηθήσει. Τώρα, στην κυρία Μονής για τις δύο πτυχές που θίξατε, τροπολογία υπάρχουν 2, για μένα είναι σαφές ότι μια αναφορά σε αυτήν τις εκλογέ δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά η δεύτερη πτυχή που αναφέρατε με την επιφύλαξη των κρατών μελών για το καθεστώς, αυτή είναι και η πρόταση του κ. Κούπερ για τον διάλογο για περιφερειακή συνεργασία και ελπίζω πως οι Σέρβοι θα το δεχτούν στο πλαίσιο του διαλόγου. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν βρίσκεται στην συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 5. Τώρα για τη συμβαστική πρόταση 6 καλωσορίζει την δήλωση του Προέδρου της ε, Σερβίας συνεργικά με την πρόταση στο, στα, στα συνεργικά σημεία ελέγχου. Ναι, περιλαμβάνεται ε, και κάτι ακόμα που θέλω να διευκρινίσω, πολλοί συνάδελφοι τόνισαν τις ανησυχίες τους και συνέψε κριτική για την ULEX. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία αναθεώρησης που συνεχίζεται και υπάρχει η ιδέα, τώρα μου αφού σας άκουσε, να υπάρξει ακρόαση με τα μέλη της CMPD και της ULEX για να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον θα προτείνω λοιπόν κάτι τέτοιο στο διευρυμένο Προεδρείο αργότερα. Να έχουμε λοιπόν μια διαδικασία στο Κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό. Ε, έγινε αναφορά επίσης στον Υπουργό Εξωτερικών του κ. Σλοβενής κ. Σπόγκερ, ο οποίος έχει οριστεί να γίνει ε, και USR και επικεφαλής του γραφείου. Αυτός ο διορισμός έγινε. Τον συνάντησα την περσμένη εδώ στις Βρυξέλλες ε, και Νομίζω ότι η επιλογή είναι, είναι σωστή και θα ξεκινήσει ελπίζω το μόνο δυνατόν να εργάζεται μόλις ε, εγκαταλείψει τη θέση του Υπουργού. Τώρα, το ζήτημα των ε, διαδηλώσεων ε, και εγώ άσκησα κριτική και θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα να οργανωθούν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους διαδηλωτές η αστυνομία ήταν και αυτός κάπως υπερβολικός, ήταν επίδειξη δύναμης. Οι διαδηλώσεις οι οποίες έγιναν χθε σε ό,τι διάβασα ε, έγιναν ε, χωρίς να προκληθούν έκτροπα. Νομίζω πως εάν η κατάσταση συνεχιστεί θα πρέπει θα το εξετάσουμε το ζήτημα ενδεχόμενα και στην Ολομέλεια να έχουμε κάποιο ψήφισμα. Ε, αλλά αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο ε, βλέπουμε το κοσμοπέδιο από το εξωτερικό, αλλά και η Σερβία επίσης. Ε, αυτά είναι ζητήματα που ήθελα να θίξω. Τέλος, να ευχαριστώ τη γραμματεία και την Εύα για την υποστήριξη της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω πως η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 9. Παρακαλώ μην ξεχάσετε τις πιστοτικές σας κάρτες. Ναι, είναι πίστος για τη δημοκρατία. Without, uh, without... Uh, Αμέσως, χωρίς να χρονοτριβήσουμε, περνάμε στο επόμενο σημείο. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την έκθεση προόδου για την πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο εισηγητής Ριχάρδος Χόουιτ θα λάβει πρώτος το λόγο. Ορίστε κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Γραμματεία πρόσθεσε το θέμα αυτό γιατί δεν είχαμε προλάβει την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ και την συνάδελφο και φίλο κυρία Λούνατσεκ. γιατί ως νέος εισηγητής θέλω να βασιστούμε και σε προηγούμενες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων. Λοιπόν, στην έκθεση αυτή θα σας επαναλάβω σύντομα τις αρχές της σύνταξής της. Ελπίζω να με υποστηρίξετε. Θέλω να είμαστε πολύ θετική ως προς την υποψηφιότητα της χώρας για ένταξη στην Ένωση και να αρχίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα οι ενταξιακές συνομιλίες όπως είπε και το Κοινοβούλιο πέρυσι. Υπήρξε καθυστέρηση και γι' αυτό χρειάζεται να δείξουμε κάποια ενθάρρυνση Γι' αυτό χρησιμοποίησα πολύ θετική γλώσσα για τα κατορθώματα της χώρας αυτής ως προς τα κριτήρια διαφανείας και λοιπά και ακόμη και για το μπάσκετ είπα θετικά λόγια. Μου λένε γιατί, μα για να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στον πληθυσμό της χώρας που θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για να ακουστούν αυτά και από το λαό. Γι' αυτό είπα για τον μπάσκετ λοιπόν. Στην παράγραφο 1 και στην πρώτη φράση ήδη λέω ρητά ότι θέλουμε να αρχίσουν οι ενταξιακές συνομιλίες. Γι' αυτό όλες τις τροπολογίες που την αφορούν τη συνεδίασα σε μία νέα παράγραφο 1α. Τώρα, Αφού στείλουμε αυτά τα ενθαρρυντικά μηνύματα, μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα και την ευκαιρία να πούμε και μερικά δύσκολα πράγματα για τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνει η χώρα αυτή. Λέω και δύσκολα πράγματα όπως για την ελευθεροτυπία, για την ανάγκη πολύ μεγαλύτερων, σοβαρότερων μέτρων για την αποκέντρωση, για την ανεξαρτησία της κοινωνίας των πολιτών, για την αστυνομική επιτήρηση. Αυτά είναι όλα δύσκολα θέματα, αλλά πιστεύω ότι αν τα συνδυάσουμε με στεναρή ενθάρρυνση θα ακουστούν οι επικρίσεις μας. Γι' αυτό θέλω πάνω απ' όλα ισορροπημένη και επικοδομητική και αντικειμενική έκθεση για να στηρίξουμε έτσι τις μεταρρυθμίσεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αφιβολίες από πολλούς. Ελπίζω όμως να συμφωνήσουν και εκείνοι ότι θέλησα να συμπεριλάβω τις περισσότερες σχεδόν όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν Μερικές βέβαια δεν μπόρεσα να τις υποστηρίξω ούτε να κάνω συμβιβασμούς, θα τις πω και αυτές. Αλλά 164 τροπολογίες, οι τροπολογίες είναι πολλές όπως καταλαβαίνετε και πιστεύω ότι η συμπερίληψή τους καταλήγει σε όντως ισορροπημένο κείμενο αφόσον στηρίζω τις περισσότερες από αυτές είτε ως έχουν είτε μέσω συμβιβασμών. Θέλω λοιπόν να υπάρξει συνένεση και ελπίζω να το πετύχω. Στα πολύ λεπτά θέματα, όπως το μηχανισμό μεσολάβηση στην παρέμφωθέκα, όπου ακούστηκαν αντιρρήσεις από τους πράσινους, ή για το θέμα του κατά πόσον η πάτη εκπρόσωπος έχει βοηθήσει ή όχι τα πράγματα. Για τα φορολογικά ο κ. Κόβατσεφ έχει καταθέσει σχετικά τροπολογίες όπως και ο κύριος Κύριλοφ και άλλοι. Για την τροπολογία 102 και τις ελληνικές τροπολογίες, για όλα αυτά συζήτησα με τους συντάκτες λέγοντας ότι να βασιστούμε στο περσινό κείμενο του Κοινοβουλίου και με βάση αυτήν να επαναδιατυπώσουμε τις τροπολογίες και αντιρρήσεις σας. Καταλαβαίνω ότι θέλετε τα θέματά σας να αναφέρονται στο κείμενο, ότι θέλετε να γίνει αυτό επειδή ακριβώς αντιπροσωπεύεται τις πολιτικές ευαισθησίες που αντιπροσωπεύεται αλλά επιμένω να επιμείνουμε σαν βάση στον περσινό συμβιβασμό. Τις προφορικές τροποποιήσεις που ζητάω τις βλέπετε στον κατάλογο. Τώρα το θέμα της ονομασίας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό αλλά βέβαια είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Όπως είπα και στις ανταλλαγές απόψεων και σε συναντήσεις με τους Κιώδης και διάφορους άλλους συναδέλφους, το θέμα αυτό θέλω να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά οι Έλληνες συνάδελφοι ήθελαν να τεθεί ευρύτερα στο θέμα των περιφερειακών αυτό δεν μπόρεσα να το πετύχω με το χρόνο που είχα. Μιλάω και για την ονομασία, αλλά με ταπεινό τρόπο. Δεν πάω τόσο μακριά όσο οι πράσινοι που κάνουν και συστάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Δεν είναι δικός μας ρόλος αυτός. Αλλά του συνόλου του Κοινοβουλίου και της Ένωσης να δώσει ενθάρρυνση για την επίλυση του θέματος, αλλά όχι να ζητήσει τη λύση ε, το ίδιο. Και υπάρχει και το πολύ αμφιλεγόμενο θέμα του τι θα κάνουμε εμείς για την ονομασία, τι θα, πώς θα ονομάσουμε τη χώρα στο κείμενο. Ξέρουμε ότι από το 1995 στον ΟΗΕ υπήρξε το όνομα ΦΥΡΟΜ και έχουμε την νομική υποχρέωση να το χρησιμοποιούμε. Αλλά θα ήθελα, συνάδελφοι, στο κοινοβούλιο μας να μην είμαστε προκλητικοί προς κανέναν ως προς την ονομασία. Και τι έκανα λοιπόν, κάθε παραπομπή στο όνομα είναι είτε Φιρόμ είτε Μακεδονία. Και το ένα και το άλλο. Ή μάλλον όχι, τα έβγαλα και το Φιρόμ και το Μακεδονία. Και χρησιμοποιώ εκφράσεις αυτή η χώρα και τέτοια για να μην πάρουμε θέση. Ο τίτλος της έκθεσης θα λέει «Φυρόμ». Είμαστε νομικώς υποχρεωμένοι αυτό το όνομα να χρησιμοποιήσουμε, αλλά προσπαθώ στο ίδιο το κείμενο να μην το συστηματοποιώ. Υπάρχει όμως μία παράγραφος όπου γίνεται η σύσταση να χρησιμοποιείται το επίθετο μακεδονικά για τη γλώσσα. Και αυτό το έκανα, όπως είπα και στις ανταλλαγές απόψεων, παίρνοντας κατά λέξη μία συμβιβαστική παράγραφο που είχε εγκριθεί από την Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή το Νοέμβριο. γιατί είχε αναγνωριστεί ότι η χώρα διαμαρτυρήθηκε όταν η Κομισιόν δεν ονόμασε τη γλώσσα μακεδονική. Ο, ο ΙΕ το κάνει. Και γι' αυτό άμα την ονομάσουμε και εμείς τη γλώσσα μακεδονική θα δείξουμε στο λαό ότι ακούμε τα αιτήματά του. Μερικοί συνάδελφοι ξέρω ότι δεν θα το δεχτούν αυτό και θα το καταψηφίσουν αλλά μόνο αυτή τη μία φορά το έχω κάνει εκεί μέσα. Θα δούμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία αύριο και στην Ολομέλεια. Δεν θέλω όμως να δοθεί μάχη για κάθε παράγραφο και τελικά να αλλοιώσουμε τελείως το κείμενο και να μην συμφωνεί κανείς με αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα μία και μόνη ψηφοφορία από την αρχή και ελπίζω να τα στηρίξετε όλα αυτά τέλος στην παράγραφο 7 για το Διεθνές Δικαστήριο πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες που έλεγαν ότι ότι τα Σκόπια κέρδισαν την υπόθεση και έχασε η Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι και οι δύο πλευρές έκαναν μεγάλη προσπάθεια να μην διχτούν προκλητικές. Ούτε τα Σκόπια υπήρξαν προκλητικά και τους συγχαίρω γι' αυτό, ούτε όμως η Ελλάδα. Γι' αυτό θα ήθελα το ίδιο να κάνουμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, να επιδείξουμε την ίδια πειθαρχία. Γι' αυτό σημειώνω την απόφαση ελπίζοντας να αποτελέσει όθηση για την επίλυση της διαφοράς. Και αυτό είναι πολύ πιο επικοδομητικός τρόπος νομίζω, αντί να βρίσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε υβριστική γλώσσα, όπως θα προτιμούσαν ίσως ορισμένοι τώρα, για λεπτομέρειες. Έχω ήδη κάνει συμβιβαστική πρόταση για την πρώτη παράγραφο. Για το θέμα του pre-screening στην Επιτροπή και στο σύνολο του Κοινοβουλίου όταν είχε έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών τους του είχα πει ότι υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν πολλές δημιουργικές λύσεις αλλά δεν ήθελα να το ζητήσω αυτό επίσημα γιατί θα ήταν υποτιμητικό. Το κείμενο λοιπόν που πρότεινα, με αυτό το πνεύμα το πρότεινα. Στην τροπολογία 25 θέλω να το καταλάβει ο συντάκτης στην παράγραφο 3. για την τροπολογία του κύριου Κάτσιν. Θα ήθελα να προσέξει ότι και στο σκεπτικό λέω ακριβώς τα ίδια. Την δέχομαι αλλά δεν τη δέχομαι ως τροπολογία εκεί που την ζητάει. Παράγραφος 4. Η κυρία Κοπά δυστυχώς δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα αλλά συζήτησα μαζί της και εξέφρασε την ιδέα να βγάλουμε τη λέξη θεμητή απογοήτευση, τη λέξη θεμητή. τουλάχιστον ως προς την ημερομηνία της έναρξης των συνομιλιών. Νομίζω ότι η πρότασή της είναι επικοδομητική και δέχομαι τη διαγραφή αυτής της λέξης και άλλες τροπολογίες της. Και αν χρειαστεί θα καταψηφίσω και ο ίδιος τη συμπερίληψη της λέξης. Για τον νέο ηγέτη της αντιπροσωπείας στην παραγραφό 5 Δεν πίστευα ότι θα υπάρξουν τόσες αντιδράσεις. Ήξερα ότι θα χρειαστεί να αλλάξει η διατύπωση μετά της, την αντικατάσταση του Προέδρου ή του ηγέτη της αντιπροσωπείας. Θα γίνει αυτό. Εγώ προτιμώ επ' αυτού την τροπολογία του ΕΛΚ. και θα την υποστηρίξω και αποσύρω τη δική μου. Δεν νομίζω όμως ότι η έκφραση ομιλίες μίσους είναι κάτι θετικό. όπως ζήτησε στην τροπολογία του κύριου Σκόβατσικ και άλλοι. Η κυρία Γιαννάκου υποστηρίζω αυτά που πρότεινε και που συστήνει για τις εκλογές. Εξήγησα ήδη στους πρασίνους ότι οι αντιδράσεις τους είναι υπερβολικές και νομίζω ότι η δική τους τροπολογία θα στείλει λανθασμένο μήνυμα και νομίζω ότι το δέχτηκαν. Τροπολογία 89 του κυρίου Ντέβα για τον κατώτατο μισθό. είναι κάτι που θα μπορούσα να το δεχτώ, αν και κάτι ανάλογο λέει και το κείμενο. 82, 52, 93, 97 και 102 Σόπφλιν και άλλων καθώς και 98 και 112 για την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και για τα νομικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην προενταξιακή περίοδο. Αυτές οι τροπολογίες είναι καλές και τις δέχομαι. Και ευχαριστώ τους συντάκτες για την ποιότητά τους. Για το δημοψήφισμα είχα εξηγήσει ήδη στον κύριο Κόβατσεκ ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα και αυτό μου είπαν και οι ίδιοι εκπρόσωποι της χώρας ή μάλλον για την απογραφή, όχι για το δημοψήφισμα, για την απογραφή. Είναι καλύτερο η απογραφή να γίνει γρήγορα παρά πιο αργά. Η χρήση όμως της λέξης ε, segregation για τις ε, εθνοτικές ομάδες είναι κάτι που είναι ίσως πολύ σκληρό και αυτό το απευθύνω στον κύριο Κάτσιν, είναι προκλητική λέξη. Μπορούμε να πούμε διαχωρισμός, κάτι πιο ήπιο, όπως separation. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Uh, ευχαριστώ, πολύ. Αλλά έχουμε άλλο ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Έχουμε 11 αγορητές, 12 όχι, είσαστε ήδη γραμμένος κύριε Τάνοκ. Παραμένουν 11. Α, και ο κύριος Βεγγίνεν. Λοιπόν, σκιώδεις οι είδες θα λάβουν το λόγο. Κύριος Κούκαν. Και παρακαλώ μην μακρηγορείτε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χαουίτ για την ε, σύνταξη της έκθεσης, τη συνεργασία και για τη λεπτομερή συζήτηση για τις τροπολογίες. Βρήκαμε νομίζω κάποιο περιθώριο συμβασμών που θα γίνουν δεκτές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Όχι πλήρως, ας είμαστε ρεαλιστές, είναι πολύ πλοκό το ζήτημα, οπότε συνένεση δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει φέτος. Στη συζήτηση για την έκθεση εγώ αναγνωρίζω την πρόοδο που σημείωσε η Υπουργού μου το τελευταίο έτος, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζω την άποψη πως σε πολλούς τομείς οι αρχές της Υπουργού θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Να τονίσω ε, κάποια ζητήματα. Στο ζήτημα έναρξης διαπραγματεύσεων συμφωνώ με τον εισηγητή και τους περισσότερους συναδέλφους πως παρά την συνεχιζόμενη συζήτηση για το ζήτημα του ονόματος, το Συμβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει τη σύσταση της Κομισιόν ε, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Εδώ πέρα έχει υπάρξει μεγάλο κενό μεταξύ του καθεστώτος υποψηφίου χώρας και της έναρξης ε, διαπραγματεύσεων. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ε, προσπάθειες ένταξης της χώρας, στην αξιοπιστία της Ένωσης και στην ε, συνολική διαδικασία ένταξη περιοχής. Ταυτόχρονα βλέπουμε πως οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ είναι το βασικό πλαίσιο για να λυθεί το ζήτημα, λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω πάντα τι σχέσει καλή γειτονία ω σημαντικό ζήτημα των διαδικασιών ένταξη. Επιπλέον, οι βασικέ προκλήσει για την χώρα παραμένουν, παραμένουν στου ε, χώρες, στους χώρους δικαιοσύνης και εσωτερικών, διαφθορά ειδικά στα υψηλότερα επίπεδα, ελευθερίας των ΜΜΕ και δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Σε όλα αυτά βλέπω την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες των αρχών της χώρας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την σημασία της κοινοβουλευτική συνεργασίας και του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ο βασικός ρόλος του Κοινοβουλίου στην πολιτική συζήτηση είναι βεβαίως κάτι το οποίο αποδέχονται όλοι. Πρέπει όμως να τονίσουμε πως θα πρέπει να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος στο Κοινοβούλιο μεταξύ των κομμάτων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό χαίρομαι για το ότι το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου το περσινό ε, έχει πλέον λήξει. Τέλο να πω πως ε, οι συμβασικές απολογίες φαίνεται πώ είναι αρκετά ισορροπημένε και τι στηρίζω. Ευχαριστώ. Νικολάη. Thank you, Chair. Uh, I want to Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συγχαρώ τον συγητή ειδικά για τις συμβαστικές τροπολογίες που συζητήσαμε. Οπωσδήποτε είναι ευαίσθητη και σημαντική αυτή η έκθεση λόγω του ζητήματος ε, που για μένα είναι ακόμα ευαίσθητο αλλά εγώ θα ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ανοιχτοί για την έναρξη δεξιακών διαπραγματεύσεων. Είναι φυσιολογικό το Συμβούλιο να ακολουθεί την σύσταση της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Το ζήτημα του ονόματος τώρα θεωρώ πως η απόφαση του, της Χάγης πρέπει να γίνει σεβαστή και οι δύο πλευρές και η Μακεδονία πρέπει να ξεκινήσει στο μοτρό δυνατόν τις διαπραγματεύσεις. Ε, υπάρχουν τώρα δύο ζητήματα που παραμένουν επίμαχα η δικαιοσύνη, δικαιώματα μειονοτήτων και η ελευθερία των ΜΜΕ. Αλλά νομίζω οι συμβαστικές τροπολογίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Τόσο στηρίζουμε εδώ πέρα την τροπολογία του Βουλγαρού συναδέλφου. Πρέπει να σεβαστούμε δηλαδή τα δικαιώματα των μειονοτήτων γιατί είναι σημαντικό ζήτημα για ολόκληρη την περιοχή γιατί υπάρχουν πολλές μειονότητες παντού στην περιοχή και αυτό είναι προαπαιτούμενο για την κατανόηση και την ειρηνική συμβίωση στην περιοχή και επίσης ε, θεωρώ πως η κατάσταση των ΜΜΕ πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις αρχές ε, γιατί ε, η διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η ελευθεροτυπία είναι κρίσιμα σημεία για την δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ. Πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την λέξη θεμητός στην συμβαστική τροπολογία 3. Η Πουγουδουμού ε, έχει τα τελευταία τρία χρόνια συμμορφωθεί με τα κριτήρια και υπάρχει η σύσταση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτές δεν ξεκινάνε όχι λόγω των κριτήριων, αλλά λόγω ενός διμερούς ζητήματος που δεν είναι κριτήριο. Οπότε θα έλεγα πως πέρα από οτιδήποτε άλλο, νομίζω πως είναι μια θεμητή απογοήτευση. Και στόχος μας είναι να πούμε πως το διμερές αυτό ζήτημα οπωσδήποτε πρέπει να ξεκαθαρίσει, να υπάρξει μια λύση. Αλλά μην το κάνετε εντός της διαδικασίας διεύρυνσης. Μην ε, δηλητηριάζετε τη διαδικασία διεύρυνσης με αυτό. Και βεβαίως ε, εξού και η ιδέα ενός μηχανισμού διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μεταξύ αυτών των δύο χωρών, αλλά υπάρχουν και πολλά διμερεί ζητήματα. Ακόμα και η Ολλανδία και η Δανία έχουν διαφωνίες για τα σύνορά τους. Αυτό νομίζω μπορεί να βοηθήσει και αυτό το διμερές ζήτημα να φύγει από την, αναπεμπλακή τη διαδικασία διεύρυνσης. Είναι σημαντικό λοιπόν μου να ξεκινήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στα διάφορα κεφάλαια. Συνολικά είμαι ικανοποιημένη με όλες τις συμβαστικέ τροπολογίες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε πει για ελευθεροτυπία, ε, αντιμετώπιση των διακρίσεων, ε, δικαιοσύνη και ελπίζω το έτος που έρχεται να έχουμε κάποια πρόοδο και να ξεκινήσουμε σας ευχαριστώ κύριε Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας και η κυρία Κορνιλέσεν. Πράγματι έχετε δίκιο, είναι μια θεμητή απογοήτευση για το κοινό της χώρας. Η Μακεδονία αυτή, όπως ξέρετε, η χώρα αυτή δεν θριαμβολόγησε όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ε, για την ένταξή της ε, στο ΝΑΤΟ και νομίζω πως η απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να αποτελέσει και προηγούμενο για την ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ε, ε, έλεγε πως έβαλαν τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω πως η έκθεση αυτή είναι πράγματι αντικειμενική για την ε, Μακεδονία η οποία είναι μια μικρή χώρα εύθραυστη. Βεβαίως οφείλω να σας πω εδώ πέρα πως ε, είμαι μέλος της ομάδας φιλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μακεδονίας και απογοητεύτηκα για το βέτο το οποίο ασκήθηκε κατά της σύστασης της Κομισιόν και εξάλλου η Μακεδονία είναι υποψήφια χώρα εδώ και 7 χρόνια και δεν νομίζω πως θα πρέπει να την μπλοκάρει ε, η Αθήνα ε, λόγω αυτής της διμερούς διαφωνίας μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων για το όνομα, η οποία είναι ακατανόητη για κάποιον τρίτο π.χ. στο μέλλον η Κροατία θα προσπαθήσει να μπλοκάρει την ένταξη της ε, Σερβίας ε, και άλλες χώρες ε, εμποδίζονται επίσης όπως το Μαυροβούνιο. Η χώρα λοιπόν αντιμετωπίζει εσωτερικές εντάσεις με κάποιες μειονότητες οι οποίες θέλουν να υπονομεύσουν την εδαφική της ακεραιότητα. Οπότε όσο γρηγορότερα ξεκινήσει οι ουσιαστική διαπραγματεύσεις για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, τόσο το καλύτερο. Και βεβαίω έτσι θα ανοίξει η πόρτα για περισσότερες άμεσε ξένες επενδύσεις, ε, αναπτυξιακές προοπτικές και περισσότερη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να ομολογήσω ότι ο εισηγητής μας, ο σημερινός εισηγητής, τόσο στην έκθεση όσο και κυρίως στην προφορική παρουσίαση που μας έκανε σήμερα, προσεγγίζει το θέμα με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το αναγνωρίζω. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και μάλιστα από την προφορική παρουσίαση κατάλαβα ότι επιχειρεί να φτιάξει και το διάλογο με έναν τρόπο ούτως ώστε να βρεθεί και λύση. Η θέση της ομάδας μας είναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και προφανώς και η Φύρων πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλός λοιπόν ο εισηγητής ενθαρρύνει και πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή την κατεύθυνση. Έστω και αν υπερβάλλουμε καμιά φορά με την ομάδα μπάσκετ και τα λοιπά φύλλα είμαι και αν το ψάχνει κανεί θα μπορεί να μην ήταν και τόσο περήφανο για αυτή την σύνθεση τη ομάδα και τα λοιπά. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που γίνεται να ενθαρρυνθούμε να δώσουμε την ενθάρρυνση. Το ερώτημα είναι αν από αυτή την ενθάρρυνση, όχι της ομάδας, τι καταλαβαίνει η ηγεσία αυτής της χώρας και λέω με την ευρύτερη έννοια. Γιατί τόσο καιρό δείχνει μια αδιαλαξία κατά την άποψή μου να προσεγγίσει το θέμα α, της ονομασίας με μια αμοιβαία λύση. Η ελληνική πλευρά την έχει κάνει το μισό της απόστασης. Και λέω διότι πρόσφατα από την ηγεσία της ΦΥΡΟΜ είχαμε μια απαξιωτική δήλωση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και με την πρωτοβουλία του κυρίου Νίμιτς. Για να μην αναφερθώ σε άλλα που φτάνουν στα όριο της γραφικότητας για να υποστηριχτούν ορισμένες απόψεις. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, επειδή το θέμα συνεχώς μας απασχολεί, <clears throat> δεν προέρχομαι από κυβερνητικό κόμμα που χειριστεί, στην Ελλάδα που έχει χειριστεί το θέμα αυτό, αλλά η αίσθηση είναι ή αν θέλετε η προσέγγιση που πρέπει να γίνεται είναι ότι δεν είναι μια αιμονή ή ένα διμερές πρόβλημα της Ελλάδας και της Φύρο. Δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα διεθνές και εφόσον βρίσκεται στο πλαίσιο του ΕΕ πρέπει να διευκολύνουμε στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αν θεωρηθεί ή όσο θεωρείται ότι είναι διμερές πρόβλημα τότε πραγματικά σου λέει άλλος είναι ακατανόητη αυτή η οσο θεωρειται οτι ειναι διμερες προβλημα τοτε πραγματικα σου λεει αλλωστε ειναι ακατανοητη αυτη η σταση Δεν είναι αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο ένα συμβολικό αγώνα, είναι μια πραγματική κατάσταση. Μακεδονία λέγεται μια ευρύτερη περιοχή που ένα κομμάτι της ανήκει στην ελληνική επικράτεια, ένα κομμάτι στη Φύρο, ένα κομμάτι εκεί. Και βεβαίως πίσω από αυτό έχουν ακουστεί, λέγονται και τα συμφραζόμενα, αμφισβητήσεις και ούτω καθεξής. Είναι έτσι λοιπόν φορτισμένο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει συμφωνία αμοιβαία αποδεκτή. Άρα η δική μας η προσπάθεια, η προσπάθεια ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη, δηλαδή τη διαδικασία συζήτησης, αναζήτησης, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στα πλαίσια του ΕΕ πρέπει να την διευκολύνει. Άλλες παράπλευρες διαδικασίες έχω πολλές αμφιβολίες αν μπορούν να βοηθήσουν. Παραδείγματο χάρη, είπε ο συνάδελφο και για ένα άλλο θέμα, είναι μια θέση αρχή βεβαίω. Δεν θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ και η συνύπαρξη στο ΝΑΤΟ θα αποτελέσει συγκολητική ουσία. Το αντίστροφο θα έλεγα είναι άλλη κουβέντα ω προ αυτό. Επομένω, η δική μα τοποθέτηση πρέπει να βοηθάει αυτό, να σπάει την αδιαλαξία, να διευκολύνει στο να βρεθεί το συντομότερο δυνατό λύση του προβλήματο, ούτω ώστε να επικεντρωθεί και η ηγεσία και ο λαό στη λύση προβλημάτων που υπάρχουν, δεν αναφέρομαι σε αυτά. Νομίζω ότι στα βασικά σημεία, δηλαδή τι μεταρρυθμίσεις, τα δημοκρατικά δικαιώματα, η έκθεση βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και επομένω αυτά τα σημεία τουλάχιστον θα τα υποστηρίξουμε. Τέλος, πάντα με αυτέ τι εκθέσει των υποδιεύρυνση, λοιπόν, ένταξη χωρών, η παρατήρηση είναι ότι <clears throat> έτσι όπως ορισμένες φορές οι εκθέσεις μας υποδεικνύουν ποια οικονομική πολιτική πρέπει να ακολουθεί, είναι τελειώνω κύριε Πρόεδρε, Ουσιαστικά είναι σαν να αντιλαμβανόμαστε ότι οι καινούργιε χώρε είναι η διεύρυνση των αγορών των ήδη χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή και ευκαιρίε για επενδύσει κερδοφόρε για αυτού που τι κάνουν και όχι για το λαό και την οικονομία τη συγκεκριμένη χώρα. Επομένω, στο συγκεκριμένο θέμα ε, δεν θα συμφωνήσω και έχουμε διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Κοβάτσεφ ή Κόβατσεκ. Για δύο λεπτά, ακόμη κι αν είναι ο Κόβατσεκ. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Θα συνεχίσω στα, στην βουλγαρική. Ευχαριστώ τον κύριο Χάουιτ για την έκθεση του και για την επικοδομητική του θέση σε αυτό το τόσο λεπτό θέμα και επειδή είναι διατεθειμένος να, για συζήτηση και έχει συζητήσει και μαζί μου η ανοχή και οι ευρωπαϊκές αρχές αντιτίθενται αυτή τη στιγμή στις εθνοτικές εντάσεις που σημειώνονται στην περιοχή και στην υποδούλωση στην νοτιοσλαβική ιδεολογία, σε μια νοτιοσλαβιστική ιδεολογία. Και εγώ συμφωνώ να προχωρήσουν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και οι διμερείς συζητήσεις. Η πρόοδος όμως προς την ένταξη θα έλυνε πολλά προβλήματα που οφείλονται σε καταστάσεις του παρελθόντος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής που συμμερίζονται κοινή ιστορία. Θα μπορούσε και το Κοινοβούλιο να κάνει κοινού εορτασμούς και λοιπά σε ιστορικές ημερομηνίες. Ελπίζω σε έναν από τους συμβιβασμούς που θα εγκριθούν να αναφέρεται αυτό, ότι είναι λυπηρό δηλαδή που δεν υπήρξε πρόοδος προς κάτι τέτοιο και ελπίζω οι Μακεδόνες γειτονέ μας να μπορέσουν και αυτοί να ξεπεράσουν τους δεσμούς του παρελθόντος. Γι' αυτό προτείνω και ελπίζω να εγκριθεί αυτό να υπάρξει ένα άνοιγμα σύντομα όλων των θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία της μακεδονικής αστυνομίας με την πρώην μυστική Ιουγκοσλαβική υπηρεσία. Ελπίζω να το δεχτεί αυτό ο κύριος Χάουιτ. Υπάρχει θέμα εδώ ελευθερία συνείδησης και της δυνατότητος του καθενός να εκφραστεί είτε είναι Βούλγαρος είτε Αλβανός είτε οτιδήποτε άλλο. Να μπορεί να πει ποια είναι η εθνοτική του ταυτότης χωρίς αυτό να, δίνει, να γίνεται λόγος διώξεων ή στις εργασιακές σχέσεις με εργοδότη, εργαζόμενο. Ξέρω ότι και στα δικαστήρια πολλές φορές έχουν ληφθεί στρεβλές αποφάσεις για τέτοιους λόγους. Η έκθεση πάντως είναι καλή και νομίζω ότι πρέπει απλώς να λάβει υπόψη της και αυτά τα στοιχεία, ώστε να μπορέσει η Μακεδονία να προοδεύσει στην οδό προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να συγχαρώ τον κύριο Χόβιτ για την έκθεσή του. Ο συνάδελφος Κόβατσεκ έθιξε τα περισσότερα από τα σημεία που ήθελα να αναφέρω στην ομιλία μου. Ξεκινώντας να πω πως η Βουλγαρία ανέκαθεν υποστήριζε την, ε, Ευρωπαϊκή, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων. Θεωρούμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην σταθερότητα μιας ασταθούς περιοχής. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος ανεκτικότητας και αλήθειας. Τονίζω την πτυχή της ε, αλήθειας. Αυτό θα είναι και θα είναι η συμμετοχή τους σε ένα εργαλείο προκειμένου να ξεπεραστούν ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα τα Δυτικά Βαλκάνια. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ένταξη της ε, Πουγουδουμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα θέλουμε να τονίσουμε ότι ε, ομιλίες ε, και λόγια μίσους θα πρέπει να αποφευθούν. Αυτές οι δηλώσεις μίσους ε, ανήκουν στο παρελθόν και τώρα αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία του λόγου, η ελευθεροτυπία είναι ζητήματα που αφορούν στο παρόν και το μέλλον. Ε, οι ηγέτες των ε, λαών αυτών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν ε, λοιπόν λόγια μίσους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σλοβενικά διότι δυστυχώς υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. η identitete, kulture, vsega, kar je s tem povezano, ti jezik je pravzaprav. Κοιτάξτε, πρόκειται για θέμα εθνική ταυτότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα μιλήσω σλοβενικά. Ε, θέλω να εκφράσω λοιπόν την ελεγγύη μου με αυτό το ζήτημα. Το γεγονό είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδο ό,τι αφορά την ονομασία τη χώρα. Ένα πρόβλημα το οποίο διαρκεί εδώ και χρόνια. Το Βελιγράδι ε, με την ε, Πρίστινα σχεδόν κατέληξαν σε πόλεμο για την διευθέτηση ε, των προβλήματος ε, της ονομασίας Μακεδονία και Ελλάδα δεν μπορούν να πράξουν το αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω και από τις δύο πλευρές να καταβάλουν προσπάθειες και να εξεύρουν ένα κοινό όνομα, μια κοινή ονομασία και το Μαύρο Βούνιο θα ξεκινήσει οι στο ε, το θέρος ε, και η Μακεδονία θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να το πράξει και αυτή. Ε, τώρα να αναφερθώ στην τροπολογία υπαριθμών 22. Ο συνάδελφος Χόβιτ ε, θεωρεί ότι χρησιμοποιώντα τον όρο segregation ε, είμαι προκλητικός και να χρησιμοποιήσουμε τον όρο διαχωρισμό διαχωρισμός των παιδιών είναι ένας όρος τεχνικής ε, φύσης, αλλά αυτός ο διαχωρισμός γίνεται μόνο και μόνο για λόγους ε, θα φιλετιστικούς ε, ή αν θέλετε για λόγους διακρίσεων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο διαχωρισμός δεν θα αποφέρει τίποτα το θετικό. Καλό θα είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε τους ε, σωστούς όρους, τους πολιτικούς όρους. Εγώ επιμένω ότι πρόκειται για segregation, για θετική διάκριση αν θέλετε. Δεν είναι τεχνική φύσης, είναι πολιτικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πέτερλε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάουιτ για τις ε, προσπάθειές του και την ευαισθησία του σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα και για τις διατυπώσεις του. Ελπίζω λοιπόν ε, να επικρατήσουν ε, να επικρατήσει αυτή η γλώσσα και στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό το οποίο είπα για το Κωσφοπέδιο ισχύει και για αυτήν τη χώρα η οποία αναμένει την έναξη διαπραγματεύσεων εδώ και καιρό η έναξη διαπραγματεύσεων θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ε, διαδικασίας ένταξης και θα είναι αυτό επιτυχία όχι μόνο για την Πουγρομό αλλά για όλους μας όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Καμιά φορά όταν διαβάζω τις εκθέσεις προόδου της ε, Πουγουδουμού έχω την εντύπωση πως ε, ασχολούμαστε με διμερεί ζητήματα και πιο πολύ με αυτή την πτυχή ασχολούμαστε παρά με την πραγματική πρόοδο. Γι' αυτό θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα την παράγραφο 9. Στην περίπτωση της Σλοβενίας και της Κροατίας ε, καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα διμερεί ζητήματα και να ασχοληθούμε με την ένταξη. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι οι Κροάτες υποστήριξαν την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάουιτ για το ότι συμπεριέλαβε την τροπολογία μου στην συμβιβαστική ε, τροπολογία 5 στην παραγράφο 7 όσον αφορά δε το επίθετο μακεδονικός. Να σας πω κάτι από το παρελθόν. Εγώ ε, κατάγομαι από την πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Σλοβενίας. Ε, η Σλοβενία αναγνώρισε την Μακεδονία υπό το συνταγματικό της όνομα ε, και όσο ήταν βεβαίως όσο ήμασταν εντός της Γιουγκοσλαβίας δεν ήταν αυτό εμπόδιο για κανέναν. Μετά υιοθετήσαμε την ευρωπαϊκή ορολογία και χρησιμοποιούσαμε και τους δύο όρους εξίσου αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε να μιλάμε για κάποιον κάπου. Κάθε ταυτότητα πρέπει να έχει ένα όνομα και νομίζω πως θα είναι ε, και σύμφωνο με τις δικές μας αρχές ε, περί ταυτότητας να σεβαστούμε αυτή την θεμελιώδη προσέγγιση. Ελπίζω η πρώτος να συνεχιστεί. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους επένους τον κύριο Χάουιτ ε, νομίζω σωματώνει αρκετά πράγματα. Θα ήθελα όμως να αναφέρω τρία ζητήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, δεν μπορούμε έτσι απλά να αγνοούμε συνθήκες. Υπάρχει μια ενδιάμεση συμφωνία και αυτή η ενδιάμεση συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεύτερον, σημαντικό, εγώ πάντα το έλεγα, να περιμένουμε την απόφαση της Χάγης. Ε, εκδόθηκε η απόφαση της Χάγης και τώρα πάλι πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω τώρα τι περιμένουμε. Εάν ήταν αντίστροφη η απόφαση, δεν θα περιμέναμε. Οπότε είμαι κάπως επιφυλακτικός. Τρίτον, η διαγραφή της λέξης μακεδονικός. Ε, προτείνω να διαβάσετε τη συμφωνία της ε, Οχρίδος που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου γίνεται λόγος για μακεδονική γλώσσα. Ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν έχω πρόβλημα να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβασμό για το όνομα του κράτους κτλ. Παρά το ότι σας είπα δεν το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν ε, περιοχές με το ίδιο όνομα και σε άλλα κράτη που γειτονεύουν και δεν οκλήκαν. Αλλά ούτως ή άλλως η συμφωνία της Χρήδος περιέχεται η λέξη μακεδονικός για την γλώσσα του σλαβικού αυτού πληθυσμού. Είναι ο επίσημος όρος. Και δεν μπορούμε να λέμε στον καθέναν πώς ε, ονομάζεται. Το όνομα του κράτους είναι κάτι εντάξει, που μπορούμε να συζητήσουμε και αυτό δύσκολο, αλλά το, ε, οι άνθρωποι, το, εάν την ακαδημία τους ή τη βιβλιοθήκη τους ονομάσουν έτσι, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να τους το σας ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ε, πρώην Δημοκρατίας της Μακεδονία το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. <clears throat> Υπάρχουν δύο τρόποι να συζητήσει κανείς τέτοια θέματα. Ο ένας είναι να δούμε τι λέει η πλειοψηφία και να περάσει το δικό της, αλλά οι αποφάσεις για το θέμα αυτό θα ληφθούν από το Συμβούλιο και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο άλλος είναι να λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι το κράτος αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει μία ψεύτικη ταυτότητα βασισμένη στην προπαγάνδα. Το πρόβλημα δεν είναι το όνομα κύριε Πρόεδρε, είναι η προπαγάνδα που απορρέει από το όνομα. Είναι οι γελιότητες που γίνονται και η αιμονή α, της ηγεσία της περιοχής αυτής. Every nation is propaganda ε, δεν είναι every nation's προπαγάνδα κύριε Πόζελ. Η προπαγάνδα φτάνει μέχρι ενό σημείου. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία, γιατί είναι υποχρεωτικό να πρέπει να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, ε, θα πρέπει νομίζω να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τα προβλήματα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω των τροπολογιών, των συμβαστικών του κυρίου εισηγητού. Η ένα, δύο και τρία για μένα δεν είναι αποδεκτές. Η τροπολογία 5 ε, δεν μπορεί να καλεί και τις δύο κυβερνήσεις να αποφύγουν επιθετικές ενέργειες, διότι οι επιθετικές ενέργειες και προπαγανδιστικές και εργαλειοποίηση της ιστορίας γίνεται από την πλευρά των Σκοπίων. Η τροπολογία 6 σχετικά με τη χρησιμοποίηση του όρου μακεδονικός φυσικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο όρος αυτός. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω κάτι. Το Κοινοβούλιο αποκαλεί τη χώρα αυτή former Yugoslavic Republic of Macedonia. Πώς κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί στην έκθεσή της δεν λέει σκέτο Μασεντόνια. Αυτά είναι ασύμβατα. Δηλαδή θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, λίγο πρέπει και εμείς οι ίδιοι ας πούμε να είμαστε συγκεκριμένοι και αληθείς. Τώρα στην τροπολογία 20, οι υπόλοιπε τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνος, στην τροπολογία 20 η συμβιβαστική δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα των τροπολογιών. Πού το βρήκε η τροπολο... ο εισηγητής ότι πρέπει να υπάρχουν ε, με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ε, κοινό, κοινός τρόπος εκπαίδευσης κτλ. Δεν γράφει πουθενά καμία τροπολογία περί Ελλάδος. Και τέλος την τροπολογία 21 κύριε Πρόεδρε, εάν δεν λυθούν τα προβλήματα που αφορούν στην απόφαση και στην συνέβρεση συμφωνίας υπό το ε, Ηνωμένα Έθνη για το όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Εγώ το έχω πει πολλές φορές εδώ, ορισμένοι θεωρούν ότι αν επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια, τελικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει όπως θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είμαι και πιο σύντομο. Πρώτα απ' όλα να πω πω ο κύριο Χάουτ προετοίμασε μια εξαιρετική έκθεση με ναι, τρόπο ανοιχτό και αξιοπρεπή. Και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η πρώτη του έκθεση για το θέμα αυτό. Ναι, είναι φυσιολογικό το ζήτημα του ονόματος να είναι το επίκεντρο των συζητήσεων, γιατί φαίνεται πως ό,τι και αν κάνουμε, πάντα εκεί πέρα κολλάμε και εμποδίζεται οποιαδήποτε άλλη πρόοδος. Δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία και τώρα ο Γκρουεύσκι πρέπει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που είναι λιγότερο διατεθειμένη για συμβασμό από την προηγούμενη. Ας έχει. Τώρα πρέπει να βρούμε μια λύση. Εγώ υποστηρίζω αυτό το οποίο λέω στην εκθεσή μας για μεγαλύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία γιατί προφανώς εάν βασιζόμαστε μόνο στον ΟΗΕ δεν, δεν έχουμε αποτελέσματα θα πρέπει ίσως να βρούμε έναν τρόπο να ενθαρρύνουμε και τις δύο χώρες να αναζητήσουν μια λύση στο ζήτημα του γονόματος. Όμως ο χρόνος περνάει και τίποτα δεν αλλάζει. Οπότε δεν θα πρέπει να είμαστε όμοιροι αυτού του διμερούς ε, ζητήματος, γιατί έτσι είναι η εσωτερική σταθερότητα της χώρας, είναι σαφές, και άρα την ε, ασφάλεια ολόκληρη περιοχή. Η Βουλγαρία ως ε, χώρα που συνορεύει πρέπει να το πει ξεκάθαρα. Οπότε δεν μπορούμε ίσως να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά μπορούμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση που να ε, δεσμεύει ε, να εντάσει τη Μακεδονία και τους πολίτες της ε, σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κοιτάξτε, βρήκαμε μια λύση για το κοσμοπέδιο, παρά το ότι πέντε χώρες δεν ε, το έχουν αναγνωρίσει. Βρήκαμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Βρήκαμε έναν τρόπο να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία. Νομίζω πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια τέτοια λύση και με την χώρα αυτή μέχρι να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα του ονόματος. Οπότε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά θα πρέπει νομίζω να επικεντρωθούμε στις επαφές μας με την Κομισιόν γιατί είναι πιο δύσκολο με το Συμβούλιο να έχει μια ενεργητική και θετική αν θέλετε ατζέντα με τη χώρα αυτή μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και στο πνεύμα της γενεοδορίας επειδή σήμερα είχαμε και εκλογές ο Ρίτσαρτ θα έχει πέντε λεπτά για να μιλήσει για να απαντήσει σε όλα αυτά. Thank you. Ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Πραγματικά χάρηκα αυτή την έκθεση. Και πραγματικά, πραγματικά ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι. Κυρία Νικολάη, εγκατέλειψε την αίθουσα, αλλά τώρα ε, τα η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου νομίζω ότι αντανακλάται στον συμβασμό. Κυρία Κορνέλισεν, άκουσα αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνω στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας ε, που είχαμε. Έχουμε όμως μια χωριστή ψηφοφορία, αν θέλετε, πάνω στο σημείο να δούμε ποια θα είναι η θέση της ε, Επιτροπής μας. Το, για το ΝΑΤΟ, κύριε Χουντή, δεν το συμπεριλάβα στο ψήφισμα. Η συνάντηση του Σικάγο και το ΝΑΤΟ είναι ημερομηνίε και συναντήσει πολύ σημαντικέ. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Απαντώ ειλικρινά και έντιμα στο το, το θέμα. Το αυτό που είπε κύριε Κόβατσοφ, ε, με στις συζητήσεις που είχαμε στα Σκόπια και επιθυμώ να συνεχίσω. Είχαμε συζητήσει το θέμα στο Στρασβούργο, είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κούκεν και περιμένω να δω την τροπολογία. Μπορεί να έχει κατατεθεί και να μην είχα την ευκαιρία να την αναγνώσω. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορούμε μαζί να βρούμε έναν κατάλληλο συμβασμό. Ναι, στην αρχική μου παρουσίαση όντως ε, το παραμέλησα το ζήτημα Θέλησα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν πέρυσι, ήθελα να συμπεριληφθούν στον έκθεση. Τώρα κυρία Νέσκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς ε, να με επικρίνει ότι κράτησα μια θέση ιδιαίτερα ελαφριά και επιπόλαιη. κύριε Κρέσκι. Δεν ε, θέλησα να πω ότι κάποιος ε, από τα μέλη της Επιτροπής θέλησαν ε, ή επιθυμούν να παραμείνουν προκλητικοί. Ναι, εγώ χρησιμοποίησα τον όρο segregation στο αρχικό έγγραφο, αλλά Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω και αυτό το οποίο εσείς πιστεύω ότι θέλετε να δείτε είναι να μην υπάρξει αυτό, η segregation, αυτή η ε, διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό το οποίο προτείνω είναι πολύ πιο ανεκτικό αν θέλετε, πολύ πιο ενδοτικό. Δεν θέλω λοιπόν ε, Μάλλον δεν ήθελα να σας προσβάλλω και να πω ότι θέλετε να είστε προκλητικός. Στην ε, παράγραφο 9 υπάρχει μια τροπολογία η οποία έφτασε με καθυστέρηση στα χέρια μου αλλά είναι δύσκολο να την αποδεχτώ εφόσον έχουμε διαπραγματευτεί τις συνδραστικές τροπολογίες. Πάντως ε, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω μετά την ανταλλαγή ε, κύριε Πόσελ, ευχαριστώ για τα λόγια σας. Συμφωνώ με τα περισσότερα των όσων είπατε. Ε, ε, μετά αυτά που είπε η κυρία Γιαννάκου είναι ε, απολύτως αντίθετα με τα λόγια του κυρίου Πόσελ του λογοθοκοπούνται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλησα να, να ζητήσω ελεύθερη ψηφοφορία για το σημείο 8. Ελπίζω η Επιτροπή μας να ε, την υπερψηφίσει. Κύριε Γιαννάκου, επαναλαμβάνω ότι υποστηρίζω πολλές τις τροπολογίες της, ε, αλλά στην συγκαστημό 20 να ξέρετε ότι αυτό είχε συμφωνηθεί λέξη προς λέξη πέρυσι στο Κοινοβούλιο. Τέλος, ευχαριστώ τον κύριο Βεκίνεν για τα λόγια του και για την υποστήριξη της εργασίας μου νομίζω ότι έχει θέσει πολύ σωστά τα ζητήματα. Εγώ ήμουν πριν από δύο εβδομάδε στη νέα κυβέρνηση, τον κύριο Δήμα και ελπίζω ότι δεν έχει ακόμα χαθεί η ευκαιρία. Αλλά έχετε δίκιο να λέτε ότι η συνέχιση του ΣΚΒΟ δεν αποτελεί επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προχωρήσουμε παρακάτω και να μην πάρουμε στο ΣΚΒΟ. Ευχαριστώ. Ε, σας υπενθυμίζω πως αύριο το πρωί στις νέα θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Και να πω κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα γραμματικό σφάλμα παράγραφο 6. Πρέπει λέμε ευκαιρίε και όχι ευκαιρία. Εντάξει, δεν αλλάζει το νόημα, αλλά θα ήθελα να κάνω αυτή την ε, ορθογραφική διόρθωση. Να ζητήσω τώρα την κυρία Νέιτς. Διότι θα περάσουμε στο σημείο 10, συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης. Να δώσω το λόγο στην κυρία Νέιτς να ε, μας παρουσιάσει το κείμενο της. Ναι, θα μιλήσω γαλλικά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Το σχέδιο αυτό σύστασης του Συμβουλίου για την υπογραφή ενός πρωτοκόλου ευρωμεσογειακού που να συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της άλλης πλευράς της Μεσογείου ή μάλλον την κάθε χώρα της Ένωσης με το Μαρόκο αφορά πιο συγκεκριμένα τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα ενωσιακά προγράμματα. Στις 20 Δεκεμβρίου το συζητήσαμε πρώτη φορά εδώ μέσα. Αύριο θα ψηφίσουμε και επειδή δεν κατετέθη ούτε μία τροπολογία μέχρι τη διορία της 10 η Ιανουαρίου, θα περιοριστώ να σας υπενθυμίσω τα βασικά. Το πρωτόκολλο αυτό, ή μάλλον η σύσταση για το πρωτόκολλο, είναι να εγκρίνει το κοινοβούλιο το πρωτόκολλο. Περί τίνος όμως πρόκειται στα πλαίσια τίθεται της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και οι διαπραγματεύσεις για την πραγματοποίηση του ή για τη σύνταξή του άρχισαν από το 7 και κατέληξαν το 10. Και μετά έγινε μία πρώτη νομοθετική πρόταση στις 10 Μαΐου του 10 που συζητήθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου του 10. Το πρωτόκολλο περιορίζεται στις βασικές αρχές της συμμετοχής του Μαρόκου και ιδιαίτερα στα εξής προγράμματα ή τομείς. Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, σε είπε, Τελωνία μέχρι το 2016, Σεζάρ δηλαδή Single European Sky κλπ και Μαρκόπουλο. Μαρκοπόλο δηλαδή. Ιδιαίτερα εξηγεί τους τρόπους και τους όρους με τους οποίους θα εφαρμοστεί η συμμετοχή του Μαρόκου σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα και τομείς. Ιδιαίτερα το θέμα της χρηματικής εισφοράς του καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης που πρέπει να προβλέπει κάθε συμφωνία μεταξύ Κομισιών εξ ονόματος της Ένωσης και Μαρόκου. Σας υπενθυμίζω ότι τώρα πέρασε ένας χρόνος από την Αραβική Άνοιξη και βλέπουμε τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα. Ξέρετε ότι στο Μαρόκο το Σύνταγμα τροποποιήθηκε μετά από δημοψήφισμα που είχε δώσει τεράστια πλειοψηφία και οι βουλευτικές εκλογές έγιναν με άμεμπτο τρόπο και το κυρίαρχο κόμμα που προέκυψε από αυτές τις εκλογές ήταν το ΠΖΔ, κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης, από που προέρχεται και ο τωρινός πρωθυπουργός. Είναι ένα θρησκευτικό αλλά μετριοπαθές κόμμα Δεν είχε βέβαια απόλυτη πλειοψηφία για να κυβερνήσει μόνο του και είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει ειλικρινείς και ανοιχτές σχέσεις με το Μαρόκο. Το πρωτόκολλο αυτό μας δίνει την ευκαιρία και στην αιτιολογική έκθεση υπενθυμίζω την ανάγκη που υπάρχει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε όλες τις πτυχές της, του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι είναι απαραίτητο όποια πολιτική εφαρμοστεί με βάση το πρωτόκολλο να ωφελεί πραγματικά τον πληθυσμό του συνόλου της Μαροκινής επικράτειας μεταξύ άλλων και τη Δυτική Σαχάρα. Δεν υπήρξαν επαναλαμβάνω τροπολογίες, γι' αυτό φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι αύριο να εγκρίνουν στην ψηφοφορία και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς ο κύριος Παντζέρη, ο Αντώνιος δηλαδή. Ευχαριστώ συντομία Πρόεδρε, διότι συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια της εισηγήτριας. Και εγώ θεωρώ πως το πρωτόκολλο αποτελεί μια πράξη στήριξης και ενθάρρυνσης ισχυρής, στεναρίς που θα πρέπει να στείλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Μαρόκο προκειμένου να εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη ξεκινήσει και να προχωρήσει περαιτέρω με νέες μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει μια ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Θα πρέπει να επιμείνουμε ειδικά μετά από τις εξελίξεις στο Μαρόκο ύστερα από τις εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να συνοδέψουμε αυτό το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου με αυτά τα λόγια διότι θεωρώ ότι στην ισχύουσα φάση θα πρέπει να επιταχύνουμε την, να επιταχυθούν μάλλον οι διαδικασίες μεταρρύθμισης στο Μαρόκο. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες, και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή και τον συναδελφό Παντζέρη αναφορικά με τη στρατηγική σημασία των σχέσεων ε, μας με το Μαρόκο ότι αυτή η σχέση τώρα θα έχει καταστεί σαφέτε, σαφέστερη μετά από το, την πνοή των ε, αλλαγών και των εξελίξεων στον ε, Αφρική και στο Μαρόκο ιδιαίτερα. Όλοι λοιπόν συμφωνούμε με αυτήν την στρατηγική σημασία που έχουν οι σχέσεις και δει η βελτίωση των σχέσεων μας με το Μαρόκο. Λοιπόν, Ευρωπαίοι και Μαροκινοί θα πρέπει να βασιστούν στις κοινές αξίες που μας διέπουν και εγώ ήμουν μεταξύ αυτών στο Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκα για την κατάσταση στην ε, Νότιο Σαχάρα διότι νοιάζομαι για το Μαρόκο. Δεν έχω τίποτα αντίον του Μαρόκου. Του, του, του Είμαι Πορτογαλίδα και το Μαρόκο είναι ο δεύτερος ε, σημαντικός γείτονάς μας ε, μετά την Ισπανία. Μας ενδιαφέρει το Μαρόκο, μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο και ως εκ τούτου ένα σοβαρό πρόβλημα δεν μπορεί να κρύβεται κάτω από το χαλί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το προηγμένο καθεστώς και οι σημαντικές αλλαγές που επεκτείνονται στο Μαρόκο θα μας δώσουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, κατάματα κατάφατσα και να τα επιλύσουμε. Αυτό λοιπόν θα αποβεί προς όφελος ε, των Μαροκινών και πέραν φυσικά και των ε, κατοίκων της ε, Νοτιού Σαχάρας. Της Δυτικής Σαχάρας, συγγνώμη. Ευχαριστώ και Σπρέντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την ευρύτατη συνένεση που υπάρχει στην Επιτροπή μας ε, αναφορικά με τη συμμετοχή του Μαρόκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε η κυρία Νέτς, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα ε, και στεναρό μήνυμα προς το Μαρόκο, ειδικά στην κυβέρνηση του Αμπτελιλάν, Επιτρέψτε μου επίση να πω ότι πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την προσέγγιση ε, Μαρόκου και την Ισίας. Συμφωνούμε λοιπόν με όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται και σε αυτές που επίκυνται τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ. Αύριο το πρωί στις 9 θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Να έχετε λοιπόν τις ε, κάρτες ε, μαζί σας και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αλμπερτίνη και το επιτελείο του για την συνεργασία του και την συντροφικότητά τους. Ευχαριστώ. Τα πούμε αύριο.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

Al Atkins 120, Kobal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 Schütz Danmark like Volker Schütz.